ich bitte Παρακαλώ τους συναδέλφους να λάβουν τις θέσεις τους. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα πάλι, γεμάτο πρόγραμμα μπροστά μας. Καλωσορίζω λοιπόν θερμά τον Δανό Υπουργό για το κλίμα, την ενέργεια και τις κατασκευές, κύριο Μάρτιν Λίντεγκάρτ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνάδελφός σας, Υπουργό για Τρόφιμα Γεωργία και Ελία, ήταν το πρωί μαζί μας. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε την παρουσίασή σας για τις ε, προτεραιότητες. της Προεδρίας. Μετά θα έχουν οι συνάδελφοι τη δυνατότητα να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους. Για να απαντήσετε εσείς και μετά θα κάνουμε ένα δεύτερο γύρο. Παρακαλώ, περιμένουμε μια δημονία να ακούσουμε την ε, ομιλία σας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που έχω την ευκαιρία να έρθω εδώ και να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Η Επιτροπή σας έχει μεγάλη φήμη, ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές ε, επιτροπές και όσον αφορά την δημόσια συζήτηση και όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Θα προσπαθήσω λοιπόν να κάνω όσο καλύτερα τη δουλειά μου μαζί σας, σε συνεργασία μαζί σας και να θέσουμε τις βάσεις για τη συνέχεια. Θέλω λοιπόν στενή συνεργασία μαζί σας και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες. Η κύρια ανησυχία των κρατών μελών και των πολιτών είναι και πολύ σωστά η κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ευρωπαϊκή οικονομία και τα δημοσιονομικά μας. Ως πολιτική λοιπόν πρέπει να δράσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη τις επόμενες χρονιές. Το σώμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεντρώνει διαφορετικέ πολιτικέ οικογένειε. Αυτό που μα ενώνει είναι η πεποίθηση ότι στον αυριανό κόσμο θα τα καταφέρουμε καλύτερα αν είμαστε μαζί παρά μόνοι μα. Η σημερινή κρίση απαιτεί ενωμένη να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τρέχουσα οικονομική κρίση θα συνεχιστεί αν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε μεταξύ άλλων και την κλιματική αλλαγή, που είναι άλλη πρόκληση που αντιμετωπίσουμε. Τα τελευταία δέκα χρόνια οι τιμές των αγαθών έχουν ε, αυξηθεί περισσότερο από ό,τι όλο τον προηγούμενο αιώνα. Ήδη από το 2008 ξέρουμε ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια οικονομική κρίση. Υπάρχει και κρίση πόρων. Υπάρχει ανάγκη για όλο και περισσότερους πόρους. Οι κλιματικές αλλαγές, η μετανάστευση είναι πράγματα τα οποία αποτελούν πρόκληση για τις κοινωνίες μας. Εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αναλάβουμε δράση θα πάμε πίσω και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των τιμών. Όπως ξέρετε, Πρόεδρε, αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο η νέα κυβέρνηση της Δανίας έχει δεσμευτεί να μειώσει κατά 40% μέχρι το 2020 τις εκπομπές της διοξιδίου του άνθρακος. Και η ενέργεια αυτή θα αντικατασταθεί από την ολική ενέργεια. Η αύξηση των τιμών έχει να κάνει με την έλλειψη των πόρων επίσης. Θέλουμε λοιπόν μια οικονομία που να βασίζεται σε χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και να βασιστούμε επίσης στην ανταγωνιστικότητά μας και να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε άλλες περιπτώσεις ε, αύξησης τιμών. Πρέπει να επενδύσουμε για το μέλλον και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά τις ε, προβλέψεις μας και τα σχέδιά μας για το 2030 και 2040. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε μια τάξη στα του οίκου μας. Αυτό ήδη ξεκινάει με τη στρατηγική του 2020. Μια πράσινη Ευρώπη είναι μια πολύ βασική ιδέα για την ε, Προεδρία μας. Παρά, μάλλον όχι παρά την οικονομική κρίση θα έλεγα, αλλά ακριβώ εξαιτία της οικονομικής κρίσης. Τι προβλέπει η ατζέντα μας. Θέλουμε να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση κατά 20% το 2020, χρησιμοποιώντας πιο αποτελεσματικά την ενέργεια. η ενέργεια μας στήγησε 450 εκατομμύρια ευρώ, μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2010. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός που πληρώνουμε για το πετρέλαιο στην Ευρώπη πέρυσι αυξήθηκε κατά 100 δις ευρώ. 450 δις ήταν. Είναι λοιπόν ε, η ώρα να φροντίσουμε για περισσότερο πράσινη πολιτική γιατί έτσι θα διασφαλίσουμε το μέλλον της Ευρώπης και να μην επενδύουμε σε πετρέλαιο το οποίο παράγεται, μάλλον το οποίο εξορίσεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο έτσι θα μπορέσει να εξοικονομήσει ενέργεια και μόνο έτσι θα εξοικονομήσει και δισεκατομμύρια, ενέργεια, ε, δισεκατομμύρια ευρώ από την ενέργεια την οποία αλλιώ εισάγει. Κάτι το οποίο βέβαια δεν βοηθάει και την οικονομική ανάκαμψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι η οδηγία που προτείνει μπορεί να σώσει δεκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Ορισμένες χώρες, ορισμένοι τομείς μπορεί να μην νιώθουν πολύ καλά για, κάποιους, για κάποια σημεία της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καταλαβαίνω τις ανησυχίες. Και καταλαβαίνω επίσης ότι η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Όμως έτσι όπως έχει η οικονομική κατάσταση σήμερα είναι πολύ βασικό για να εκπονήσουμε τις πολιτικές μας, να λάβουμε υπόψη μας την εξοικονόμηση της ενέργειας. Πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές και αυτό πρέπει να φαίνεται στην οδηγία. Και ό,τι απόφαση ληφθεί πρέπει και να τηρηθεί. Αν δεν μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, τότε έχουμε πολλά να χάσουμε. Τώρα σε σχέση με την οδηγία αυτή και τις εκπομπές. Υπάρχουν και οι προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι πρώτα απ' όλα να εγκριθεί η οδηγία αυτή και είναι και προσδοκία της ε, Δανέζικης Προεδρίας. Και αυτό το έχουμε ξαναμπεί και έχουμε ευχαριστήσει γι' αυτό και τον Πίτε Λίζε και την Επιτροπή σας. Έπειτα έχουμε και την προοπτική του 2050. Έχω διαβάσει την σχετική σας έκθεση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το έχω ήδη συζητήσει το θέμα με ορισμένου από εσά, αλλά και με άλλους. Η συζήτηση αυτή είναι κλειδί για το μέλλον της μελλοντική κλιματικής αλλαγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε κάπου και θα υιοθετήσουμε τα συμπεράσματα ε, στο Συμβούλιο τον ε, Μάρτιο, φαντάζομαι. Η φωνή του δικού σας του σώματος βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Οι τιμές έτσι όπως έχουν σήμερα δεν βοηθούν στο να καταλήξουμε σε ένα χαμηλότερο αποτύπωμα η Επιτροπή σας επίσης έχει ασχοληθεί και με το θέμα του παγώματος γεών. Προκειμένου και αυτό να βοηθήσει για λιγότερη ρήπαση της ατμόσφαιρας. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίσει με την πρότασή του, τότε θα αποτελέσει η πρόταση αυτή ε, σημείο διαπραγμάτευσης στο Συμβούλιο. Το θέμα δεν είναι το αν, το θέμα είναι το πώς θα διασφαλίσουμε τις βιώσιμες πηγές ενέργειας. Μόνο λίγες ε, χώρες ε, προτείνουν μικρότερο ποσοστό για το 2030. Συνεπώς, ο ακρογωνίος λίθος του 2030 πρέπει να ισχύσει και να αποφύγουμε στραβές και λανθασμένες επενδύσεις που δεν μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Όσον αφορά τώρα το αποτέλεσμα COP17 στον Τέρμπεν, Ήταν κατά πάσα πιθανότητα ότι καλύτερο μπορούσαμε να πετύχουμε χάρη στην συνεργασία που είχαμε με διάφορες χώρες, περισσότερο ή λιγότερο αναπτυγμένες, Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τόσους πολλούς από εσάς παρόντες στο Ντέρμπαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να πιστεύει στη διαδικασία των, τρίων, των C. Θέλουμε όλες οι πλευρές να συνεισφέρουν στην ε, μείωση των κλιματικών αλλαγών. Η διπλωματία του κλίματος είναι κάτι στο οποίο δίνουμε μεγάλη σημασία και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει να μειωθεί και η οικονομική κρίση. Ορισμένοι από εμά ε, βέβαια ε, μίλησαν για τη δύναμη που μπορεί να έχει η Ευρώπη στην παγκόσμια σκηνή και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Όλοι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε μετά από τα επιτεύγματα αυτά στο Ντέρμπαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει σημαντικό ρόλο και στην συνεργασία με διάφορες αναπτυσσόμενες χώρες. Τα αποτελέσματα του Ντέρμπαν δεν φτάνουν από μόνα τους. Πρέπει να καλυφθεί το κενό μέχρι το 2020 και να φροντίσουμε να είναι αρκετά ισχυρός ο εξοπλισμός που θέλουμε να έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τότε. Ελπίζω ότι εσείς θα βοηθήσετε να ακουστεί ακόμα πιο πολύ η φωνή της Ευρώπης μετά το Ντέρμπιν, οι ευρωπαϊκές, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, συνεχίζουν και κάνουν ε, πιο εντατικέ ακόμα τις προσπάθειές τους. Ελπίζω ότι μακροπρόθεσμα θα έχουμε μια δεσμευτική συμφωνία που θα καλύπτει όλες τις χώρες για το 2020. Όμως, είναι ξεκάθαρο ότι το COP17 δεν βοήθησε να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της πρέπει να συνεχίσουν να πιέζουν τις λιγότερο φιλόδοξες χώρες, έτσι ώστε και αυτές να μειώσουν ε, τις εκπομπές τους διοξιδίου του άνθρακα. Σε σχέση τώρα με τη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, δεν έχουμε εμείς πλαίσιο για μετά το 2012. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να πετύχουν συμφωνία για τους σχετικούς κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να βασιστεί στη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών για να κάνει προτάσεις και να επιτευθούν έτσι οι στόχοι για το 2020. Στην ομάδα εργασίας εμείς θα ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, εφόσον έχει υποβληθεί βέβαια η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Κοινοβούλιο εκ παραλίλου θα αναλάβει και αυτό τις δραστηριότητές του για να σχολιάσει και να αποφασίσει για την πρόταση αυτή. Σε συνεργασία, ελπίζω. Ο κανονισμός για τα αέρια του θερμοκηπίου πάντως προσπαθεί επίσης να μειώσει τις κλιματικές αλλαγές γίνεται μια εντατική δουλειά στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και ελπίζω ότι θα πετύχουμε συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσα στην χρονιά. Είναι τεράστια δουλειά. Ελπίζουμε να καταλήξουμε σε κοινή θέση και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει η συνεργασία μας με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Είναι στοιχείο κλειδί αυτό, να συζητήσουμε νέους ε, βιώσιμους στόχους. Ξέρω ότι αύριο θα συναντηθείτε και με τον Δανό Υπουργό Περιβάλλοντος, ο οποίος και αυτός θα σας μιλήσει γι' αυτό. Υπάρχει θέμα βιωσιμότητας. Ξέρω ότι πολλοί από εσά συμφωνείτε με αυτό και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πιέσουμε διαπραγματεύσεις. Όπως ξέρετε, εξαρτώμεθα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει πρώτα να έχουμε αυτή. Επίσης, όσον αφορά τις επιχειρήσεις ε, offshore, υπάρχει κατακαιρματισμός στην ομοθεσία των κρατών μελών όσον αφορά τις δραστηριότητε offshore δεδομένης καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού πρέπει οπωσδήποτε να μειώσουμε ε, τις πιθανότητες ε, κινδύνου για αντίστοιχα ατυχήματα και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε εφόσον αυτά συμβούν. Χρειάζεται χρόνος βέβαια για την σημαντική αυτή πρόταση και σίγουρα εμείς θα παρακολουθήσουμε και το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση αυτή της Κομισιόν. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω ό,τι ερωτήσεις έχετε και για να συζητήσω μαζί σας όλα αυτά τα ζητήματα σε μια τόσο κρίσιμη για όλους ε, συγκυρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση. Είναι πολύ ευρύ και φιλόδοξο το σχέδιό σας, το πρόγραμμά σας. Ας ακούσουμε τώρα τους συναδέλφους. Κύριε Γκαρτίνη πρώτα. Ελιζαμπέτα, μέρος του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για αυτή την συνάντηση, για αυτό το ωραία σχεδιασμένο και πρέπει να πω και πιστικό πρόγραμμα. Βρισκόμαστε σε μια πολύ λεπτή και ιδιαίτερη φάση. Επιστρέφομαι από την διάσκεψη του Ντέρμπαν με αποτελέσματα τα οποία είναι αφήσιμα. Κάποιοι τα είδαν ε, με απογοήτευση και ακούστηκαν και αρκετέ επικρίσεις. Εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι δεν είμαι τόσο απεσιόδοξη, διότι Στην Ιταλία, στην ε, παράδοση την, ε, του Λαϊκού Κόμματος υπάρχουν ρητά που λένε ότι το καλύτερο είναι το εχθρό του καλού, ο εχθρός του καλού ε, και ότι, εν πάση περιπτώσει, πάντοτε αναζητούμε την ουτοπία και ότι θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση αντίθετα πιο συγκεκριμένη για να έχουμε και πιο συγκεκριμένα και από τα αποτελέσματα και να δώσουμε κάτι καλό στους ε, συμπολίτες μας γιατί, αυτή την, ε, γιατί στη σήμερα ημέρα δεν περιμένουν το τέλειο, περιμένουν κάτι όμως καλό. Ε, όμως θα ήθελα να σας πω ότι επειδή ένα από τα αδύναμα σημεία σε σχέση με την ισχυρή ε, ηγετική θέση που κρατάει η Ευρώπη στον κόσμο, υπήρξε εδώ ίσως μια έλλειψη διαφάνειας, μια έλλειψη επικοινωνίας ε, για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και ως προς αυτή την έννοια ε, θεωρώ θετική την πρόταση κανονισμού της Κομισιόν ακριβώς για το μηχανισμό παρακολούθησης και επικοινωνίας στις εκπομπές αερίων ε, του θερμοκηπίου και σε σχέση με ε, τα άλλα αέρια που συμβάλλουν στις κλιματικές αλλαγές. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς ε, σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα το οποίο εγώ θεωρώ πολύ κρίσιμο σε σχέση με την αξιοπιστία που πρέπει να έχει η Ευρώπη απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, τα στοιχεία μας που είναι συχνά και αντικείμενα ε, συγκρούσεων και να είμαστε διαφανείς και συγκεκριμένοι στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτό είναι πολύ λεπτό ζήτημα στη στιγμή που στην ουσία αντιστρέφεται η παγκόσμια γεωπολιτική και ήταν ένα από τα βασικά πορίσματα που προέκυψαν από τη συμφωνία του Ντέρμπαν, όχι πια με τη φωτογραφία της δεκαετίας του 90 με τις αναπτυσσόμενες χώρες που πια έχουν αναπτυχθεί, έχουν αναδυθεί και δεν μπορούν ε, να βρίσκονται ουραγοί ενώ έχουμε χώρες που βρίσκονται σε πιο δύσκολη κατάσταση. Το 2050, 19 χώρες που θα είναι πρώτες στην παγκόσμια οικονομία θα είναι, είναι αυτή τη στιγμή ακόμα αναπτυσσόμενες. Ε, επειδή τον Μάιο λοιπόν ήδη θα πρέπει να πάνε στο Κιώτο με δεσμεύσεις που θα αναλάβουν κάτι το οποίο πέφτει στη δικιά σας προεδρία. Πώς ε, έχετε σκεφτεί να δράσετε σε αυτή την πολύ λεπτή και σημαντική στιγμή της προεδρίας σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάινεν, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ Λίντεγκάρντ. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας. Ε, έχετε ευρία, τυχάνετε ευρίας αποδοχής εδώ στην Επιτροπή μας. Εξηγήσατε τους στόχους σας και τη Δευτέρα και όλα θα είναι η επόμενη διάσκεψη κορυφής που θα αποφασίσει για το φορολογικό δημοσιονομικό σύμφωνο. Ε, ένα οικονομικό πρόγραμμα. Ερώτησή μου λοιπόν, η Προεδρία σας θα κάνει προτάσεις για το πώς μπορούν να δημιουργηθούν πόροι στην Ευρώπη για ένα πρόγραμμα πράσινης ανάπτυξης, γιατί στις, χώρε χώρες όπου γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ύφεση, η προστασία του περιβάλλοντος και η έρευνα στην ενέργεια θα είναι λύση, θα είναι διέξοδος για την κρίση. Εμεί είχαμε προτείνει 1,2 δι για να υπάρξουν περισσότερες επιστοποιήσεις μέσα στο πλαίσιο του συστήματος των εκπομπών. Εσείς ακολουθείτε αυτόν τον δρόμο με την ιδέα προσαρμογής ενός συστήματος μέσα στο σύστημα ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από την κατάσταση αυτή όπου η τιμή του, α, του διοξιδίου του άνθρακα δεν ε, αποδίδει αρκετά χρήματα για να αποφιερωθούν στην έρευνα. Τώρα για την βιοπικιλότητα γίνεται λόγος για το 2030-40. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο στόχος για, τη δεκαετία, για το 2030, ώστε τουλάχιστον οι επενδυτές να μπορούν να ξέρουν πού πρέπει να στραφούν. Ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την ενεργειακή επάρκεια μας ικανοποίησαν αυτά που είπατε Έχω προετοιμάσει μια έκθεση καλή, αλλά δεν οφείλεται μόνο σε μένα, αλλά και στη συνεργασία των συναδέλφων. Ναι, χτες ε, αποφασίστηκε το εμπάργο κατά του Ιράν. Άρα η κατάσταση στην ενέργεια γίνεται ακόμα πιο επίγουσα Πώς θα μπορέσουμε να δράσουμε λοιπόν και τι είδου ενέργειες θα μπορούσαμε να αναλάβουμε. Εσείς ε, μιλάτε για απόδοση και επάρκεια στην ενέργεια, αλλά άλλα κράτη μιλάνε για άλλα πράγματα. Θα πρέπει ωστόσο κάποια στιγμή να αποφασίσουμε. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας αξιολόγηση. Και θα ήθελα να έχουμε στόχους και λιγότερο δεσμευτικά τα μέτρα, τουλάχιστον να είναι με τη μορφή των συστάσεων. Φαίνεται ότι μόνο η Δανία το επιθυμεί αυτό. Μήπως λοιπόν αυτό είναι λάθο δρόμο εν τέλει, το να υποστηρίξει μια διαθέση που δεν υποστηρίζει κανείς άλλος. Πάντως θα ήταν ε, μάλλον πιο εύκολα, ενδεχομένως, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να καθέται πιο δύσκολη η λήψη απόφαση. Για το ETS ε συμφωνούμε εν γέρη με αυτά που είπε ο Γιολάιρ, αλλά θα νομίζουμε ότι θα πρέπει πάνω απ' όλα να δώσουμε κίνητρα, όχι μόνο να επιβάλλουμε διατάξεις μέσω ενό ε, συστήματος ε, με κανονισμό. Να δώσουμε κίνητρα και να προχωρήσουμε με τρόπο οργανωμένο και προγραμματισμένο. Με κίνητρα 30 ευρώ, ξεκινήσαμε 70 ευρώ. Μπορούμε να βρούμε πιστεύω μια κοινή λύση και ίσως θα μπορούσατε να πείσετε τους ε, συναδέλφους στο Συμβούλιο ότι μπορούμε σε κάτι να καταλήξουμε εν τέλει με το ETS. Για το κλίμα, κλιματικές αλλαγές 2020 και υποστήριξη για το στόχο του 30%. Νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να βρεθεί συμβασμός, συμβαστική λύση. Δεν μπορούμε ακόμα να περάσουμε 5-10 χρόνια σε με το 20-30%. Στον Τέρμαν κάτι καταφέραμε, όχι όμως αρκετά. Όχι όμως όλα αυτά που θέλαμε. Και ήταν καλό να κάνουμε μια μικρή προσπάθεια για να προχωρήσουμε, για να κλείσουμε πλέον αυτή τη μεγάλη διαβάγη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μακέι, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε σήμερα εδώ. Μα παρουσιάσετε τι θέσει σα για τι κλιματικέ αλλαγέ. Εδώ είμαι, με βλέπετε. Ξέρω βέβαια ότι το ζήτημα των αερίων σχιστολιθικού πετρώματος και σχετικής παραγωγής έχει πολλά δυσκολίες δεις και σε επίπεδο συμβουλίου. Θα πρέπει, πιστεύω, να προχωρήσουμε. Ξέρουμε ότι έχουν ε, καθυστερήσει οι αποφάσεις του Συμβουλίου, μάλλον συζητήσεις του Συμβουλίου, γιατί δεν είναι σε θέση το Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις. Πάντως το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει την Επιτροπή Χιντεργκάρτ μέχρι τώρα στις θέσεις που έχει εκφράσει όταν λέει ότι θα πρέπει η οδηγία για την ποιότητα των ε, καυσίμων να αντικατοπτρίζει και την πραγματικότητα σε σχέση με τα όσα γνωρίζουμε για τα καύσιμα αυτά, για τα καύσιμα που έρχονται από... για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν ίσως μπορέσουμε να βρούμε λύσεις οι οποίες χωρίς να μας ε, κάνουν να αποκλίνουμε από, τις, ε, για τους στόχους μας για, το, για τις κλιματικές αλλαγές, να μην εξυπηρετούν μόνο ξένες χώρες. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Χιλακάκης. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ξεκινήσω με τον Τουρμπάν. όπου βέβαια έκανε καλή δουλειά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, πολλά θα είχαμε επιτύχει περισσότερα αν είχαμε κάνει τις συμμαχίες μας ε, με άλλες χώρες, μικρές ε, και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στην Δανία το 2009, θα είχαμε προχωρήσει δηλαδή πολύ γρηγορότερα αν το είχαμε επιτύχει αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως έχουμε κάποιες ελπίδες αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να προσπαθήσουμε και μόνο μου ότι η πολιτική μας για το κλίμα υπάρχει κίνδυνος να αποτύχει. Φανταστείτε να εκλεγεί ε, ρεπουμπλικανός πρόεδρος στις ΗΠΑ ε, του, του χρόνου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια τι θα γίνει τότε η προσπάθεια για την κλιματική αλλαγή. Επομένω θα έπρεπε να έχουμε μια εναλλακτική. Εναλλακτική, εάν κάτι δεν πάει καλά, εάν δεν επιτύχουν οι προσπάθειες του Ντέρμπαν και οι λοιπές διεθνείς προσπάθειες, να έχουμε μια εναλλακτική. Και έτσι περνάω στο ETS και την αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας, που είναι προφανές ότι θα πρέπει βεβαίως ε, να είχε γίνει προσπάθεια ήδη και θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με μεγάλη αποτελεσματικότητα και μόχθο. Για το ETS όμως πιστεύω θα πρέπει να το αναθεωρήσουμε. Αναφέρεστε στην ε, ε, μιλάτε για τα 7 ευρώ ως τιμή άνθρακα. Ε, σε ένα βαθμό αυτό το ορίζει το κέρδος. Σε ένα βαθμό το οφείλουμε στην ύφεση και τις οικονομικές συνθήκες σε διάφορα κράτη, σε αρκετά κράτη, που δεν επιτρέπουν, που δεν ε, ήταν δυνατόν να προβλεφθούν τρόπον τεινά. Άρα θα πρέπει να φροντίζουμε ό,τι εισάγουμε να είναι πολύ προσεκτικά μελετημένο. και να μην χρειαστεί οι χώρε αυτέ που είναι ήδη επιβαρημένε να επιβαρυνθούν με ακόμη περισσότερε, ακόμη πιο ακριβέ μέσα από το διοξίδιο, με το σύστημα των ανταλλαγών. Δεδομένου δε ότι παράγουμε και λιγότερο πολλέ φορέ στην Ευρώπη πλέον, έχουμε λιγότερη παραγωγή και ρηπαίνουμε το περιβάλλον λιγότερο εμεί, ενώ οι Κινέζοι ρηπαίνουν περισσότερο και μάλιστα και η Τουρκία γιατί είμαστε πρόσφατα στην αντιπροσωπεία εκεί και η Τουρκία προβλέπεται ότι θα έχει καλύψει την ε, κατακεφαλήν, ε, το κατακεφαλήν ποσοστό ρήπανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη στις ε, στάσεις μας, στην πολιτική που θα χαράξουμε για την ενεργειακή πολιτική και για το κλίμα βέβαια. Από την άλλη βεβαίω είναι καλό να στηρίζουμε τις θέσεις εργασίας για την ενέργεια, αλλά η θέση εργασία είτε πρόκειται για ηλιακέ κυψέλες, είτε πρόκειται για τις θέσει εργασία από τις ανεμογεννήτριες που έχετε εσεί στη Δανία, βασικά λόγω των πιέσεων τη Κίνα προέρχονται και προσπαθούμε εμείς να ε, κάνουμε τους Κινέζου να επιδοτήσουν αυτές τις θέσει. Για τις ηλιακές ε, κυψέλες ε, και τις ανεμογεννήτριες. Πρέπει λοιπόν πιστεύω με πολύ μεγάλη προσοχή να αναλύσουμε τα λάθη μας και βέβαια να τα αποφύγουμε. Ευχαριστώ πολύ λίγο ο Πρόεδρος. Αϊχάρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν στον Έλληνα συνάδελφο να πω ότι αν η Τουρκία μπει στην Ένωση θα είναι και εκείνη μέρος του, Ευρω... του συστήματος ανταλλαγής εκπομπών και θα χρειαστεί να πληρώσει. Και εκείνη, ίσως να χρειαστεί και να αλλάξετε λοιπόν θέση. <clears throat> Τώρα θα πρέπει να μιλήσω προς τον Υπουργό. Έπρεπε όμως να κάνω αυτό το σχόλιο. Επιπλέον, ε, λοιπόν, ε, ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είμαι ευτυχής που βλέπω πως έχουμε έναν φιλόδοξο Υπουργό Κλίματος ε, στην Προεδρία, γιατί το προηγούμενο μισό του χρόνου δεν είχαμε Υπουργό Κλίματος καν. Οπότε, κατά αυτή την έννοια, είναι βελτίωση. Τώρα, αν διαβάσω τα πολύ σημαντικά θέματα, είναι η επάρκεια στην ενέργεια, η διεθνή αξιοπιστία με βάση την συμμαχία που ξεκίνησε στον Τέρμπαν. Επίση, ε, ο δικό χάρτη για χαμηλό λί κατανάλωση άνθρακα. Σε αυτέ τι προτεραιότητε όλοι συμφωνούμε. Πάντω, έχω ακόμα την αίσθηση πω υπάρχουν κάποιε ασάφειε στο πώ αυτά όλα θα μεταφραστούν σε πραγματική σε, σε συγκεκριμένε δράσει. Γιατί όλα είναι αλληλένδετα. Όπω είδαμε χτε, ε, για παράδειγμα, στη, η G77 ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τις φιλοδοξίες της κλιματικής, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αν θέλουμε να βασιστούμε σε αυτή την ε, συμμαχία, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εσωτερικά. Αλλά μιλάτε και για ορόσημα στον οδικό χάρτη. Εντάξει, εφήβραμε αυτή τη λέξη milestones, ορόσημα, γιατί δεν μας άρεσε η λέξη target, στόχοι. Πάντως το ένα ορόσημο είναι 20, 2020 για 25% εσωτερικής μείωσης. Αυτό λοιπόν το διατηρούμε ως στόχο. Εκεί ήσασταν κάπως αόριστος για την επάρκεια σε ενέργεια. Όλοι ξέρουμε ότι αν θέλουμε επιτέλους να έχουμε μεγαλύτερη επάρκεια σε ενέργεια, τώρα βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει ακόμα περισσότερο πλεόνασμα ποσοστώσεων στο σύστημα ETS. Ε Τέσσερα δις ανέφερε ο Λάινεν, αλλά κάποια άλλα έγγραφα της Κομισιόν μιλάνε για 2,5 δις ε, πλεόνασμα ποσοστώσεων και οι τιμές και η Deutsche Bank, εγώ είμαι πράσινος και συνήθως δεν αναφέρομαι στην Deutsche Bank, αλλά ας το κάνω αυτή τη φορά. Λέει λοιπόν η Deutsche Bank ότι σύμφωνα με τη δική τους ανάλυση υπάρχει κρίση στον άνθρακα γιατί οι αγορές περιμένουν οι πολιτικοί να κάνουν κάτι για το ETS και γι' αυτό υπάρχει αυτή η τιμή. Και είπατε λοιπόν ναι πρέπει κάτι να κάνουμε για το ETS αλλά δεν ήταν ξεκάθαρο. Τι θα κάνουμε. Η τρίτη φάση ξεκινά στον Ιανουάριο του 2013. Οπότε το παράθυρο της ευκαιρίας για να κάνουμε κάτι είναι τώρα, στη δική σας Προεδρία. Πολύ συγκεκριμένα θα προτείνετε την... Το, να μείνουν στην, στην, στην άκρη που ε, το υποστηρίζει το κοινοβούλιο αυτό. Εμείς το υποστηρίζουμε να αναλάβετε δράση εκεί. Μπορείτε να το κάνετε με το Συμβούλιο τώρα μαζί με την Κομισιόν. Πιέστε πριν αρχίσει η τρίτη φάση. Και τέλος για να προ... κλείσουμε πρόεδρε για την ασφαλτούχο άμμο να δούμε ποιες χώρες κάνουν το δύσκολο. Η Shell, η BP, η Total, Ολλανδία, Γαλλία, Βρετανία. Αυτές μας διακυβερνούν οι εταιρείε πετρελαίου ή οι κυβερνήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε τώρα τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων και να ακούσουμε τις απαντήσεις του Υπουργού στις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ θερμά για τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Και ελπίζω ότι θα είμαι σε θέση να απαντήσω τα περισσότερα. Αλλά πάντως θα προσπαθήσω να είμαι στο δυνατόν πιο συγκεκριμένος. Πρώτα απ' όλα ο μηχανισμός ε, παρακολούθησης. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι έχει τεράστια σημασία. Όχι μόνο γιατί πρέπει να γνωρίζουμε τι κάνουμε, αλλά και γιατί είναι πολύ σημαντικό για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις άλλες μικρές χώρες. Του είπε και ο κύριος Σάικχαουτ, έχει σημασία το τι κάνουμε και τη χρηματοδότησή μας και τα αποτελέσματα που μπορούμε να περιμένουμε από, τις, ε, από τους πόρους που αποδίδουμε, που επενδύουμε και τελικά τα καλύτερα αποτελέσματα που μπορούμε να περιμένουμε. Έχει ξεκινήσει μόλις η δουλειά αυτή. Ίσως είναι μάλλον νωρίς να δώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για το φάκελο αυτό, αλλά πάντως μπορούμε να έχουμε, πιστεύω μέχρι το τέλος του χρόνου να σας δώσουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, πριν να τελειώσει δηλαδή η Προεδρία, μέχρι το τέλος της θητείας της, ε, εξαμήνου μας. Για τον κύριο Λάινεν και το σύστημα των ανταλλαγών. Ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματα του Δεκέμβριο του 2011 μας κάλεσε όλους να ολοκληρώσουμε την δουλειά ως προς την οδηγία για την αποτελεσματικότητα στην ενέργεια για να περάσουμε στο δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί εάν κοιτάξουμε τώρα το τι προβλέπει αυτή η οδηγία, εφόσον αρχίσει να εφαρμόζεται, θα φέρει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια στην ε, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ενέργειας και αυτό σημαίνει ουσιαστικό πρασίνισμα. Το Συμβούλιο λοιπόν ρητά μας ζήτησε να σημειώσουμε πρόοδο ως προς το EED, Energy Efficiency Directive. Και βεβαίως πολλοί ζητήσατε να ασχοληθούμε και με το θέμα της τιμολόγησης για να είναι σαφής η τιμολόγηση. Θα είμαι λοιπόν σαφής. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει πως ε, οι τιμές του διοξιδίου του άνθρακα είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι προβλεπόταν όταν θεσπίστηκε το σύστημα των ανταλλαγών ETS. Δεν ε, είναι βιώσιμες δηλαδή οι χαμηλές τιμές που έχουμε τώρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις τιμές στην αγορά του διοξιδίου. Ε, και πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε υψηλότερε τιμέ θεωρούμε ότι το να καταλήξουμε σε έναν οδικό χάρτη για το να άνθρακα θα, θα σήμαινε πως μπορούμε το 2030 να περιμένουμε την εξασφάλιση του στόχου του 40% και για το 2040 ακόμα περισσότερη μείωση. Θα μου πείτε βέβαια το 2020 τι γίνεται γιατί όλοι περιμένουμε βέβαια τώρα να δούμε τι ανάλυση της κατάστασης των κρατών μελών θα διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να την αναλύσουμε, να την εξετάσει το Συμβούλιο, όπως φαντάζομαι ότι και εσείς θα συζητήσετε. Επίσης, και όπως γνωρίζετε, η κατάσταση στο Συμβούλιο είναι εξή. Τρεις χώρες, Δανία, Ενωμένο Βασίλειο, Σουηδία, υποστηρίζουν να ανεβάσουμε την υποχρέωση μέχρι το 30%. Εάν όμως δεν υποστηρίξει το Συμβούλιο, εάν δεν πιεστούν ή δεν πιέσουν τα ίδια τα, άλλα κράτη-μέλη, ε, και θα ήθελα βεβαίως και να πω ότι και εσείς όσο θα πρέπει να πιέσετε, γιατί ξέρω ότι θέλετε τον ε, πιο υψηλό στόχο, τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να επιτύχουμε το στόχο του 30% το, του 20% για το 2020. Αυτά λοιπόν. Άλλο θέμα είναι αυτό της αγρανάβωσης ή της ε, διακοπής χρήσης. Θα κοιτάξουμε τα συμπεράσματα, θα επιδιώξουμε συμπεράσματα για τον οδικό χάρτη. Θα κοιτάξουμε να περάσουμε το θέμα της ε, ε οδηγίας για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα το έχετε δυνατό το αργότερο πριν το τέλος της, της ε, Προεδρίας μας και πάντως επίσης το θέμα του ε, άνθρακα και των ανταλλαγών, του συστήματος ανταλλαγών. Θέλουμε να τα κοιτάξουμε όλα αυτά τα θέματα λοιπόν, αλλά με τη σειρά το καθένα, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να περιγραφούμε σε σύγχυση να τα μπερδέψουμε, αν τα μπερδέψουμε όλα μεταξύ του. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση για το ETS φέτο, αλλά ίσω να μπορέσουμε να το κλείσουμε φέτο. γιατί δεν έχω αρκετό, ίσως δεν έχουμε αρκετό χρόνο γι' αυτό. Αλλά ίσω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Και τώρα, ο Πέτερ Λίζα. Ναι, πρέπει να ξανακοιτάξω για να θυμηθώ όλες τις ερωτήσεις. Ήταν όλες πολύ καλές. Δεσμευτική στόχη. Μάλιστα. Ναι, Τη οδηγία. Κάναμε συζήτηση στο Συμβούλιο πριν από χρόνια. Ε, λέγαμε ότι θέλαμε δεσμευτικούς ε, κανόνες ε, για τα κράτη-μέλη και κάποιες ενδείξεις για το πώς θα τους επιτύχουν, πώς θα επιτύχουν δηλαδή τους ε, ε, στόχους αυτούς του μυστικούς στα κράτη-μέλη. Εγώ προς το παρόν δεν βλέπω κάποια αλλαγή στην κατάσταση του Συμβούλιο ώστε να πω ότι έχει αλλάξει κάτι και ως εκ τούτου νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτά που έχουμε. Η πρόταση του Κοινοβουλίου τώρα, της Επιτροπής, της Επιτροπής Βιομηχανίας δηλαδή, ε, πιστεύω ότι με αυτό το δεδομένο, σε αυτό το δεδομένο στηρίζεται. Η Δανία, η Προεδρία της Δανίας, βεβαίως και μπορεί να είναι ευέλικτη ως προς το πώς θέλουμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, αυτό είναι το βασικό. Και ο μόνος τομέας στον οποίο δεν μπορούμε να, δώσουμε, να δείξουμε ευελιξία είναι ότι πρέπει να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, να ικανοποιήσουμε τους στόχους, να τηρήσουμε τους στόχους που έχει ορίσει το ίδιο το ε, Συμβούλιο. Αυτό είναι όλο. Το πώς θα το επιτύχουμε είναι μια άλλη ιστορία. Ελπίζω λοιπόν να τα καταφέρουμε. Επίσης μια πρόταση οδηγίας ε, για τα, τις εκπομπές ε, θερμοκηπίου σε διάφορα είδη καυσίμων. Από ό,τι ξέρω, συζητείτε ακόμη στην λεγόμενη Επιτροπή Ποιότητας Καυσίμων του Συμβουλίου. Ελπίζω, όπως φαντάζομαι και εσείς, ότι έχουμε κάποια πρόοδο ή θα έχουμε κάποια πρόοδο σχετικά σύντομα και ότι θα βρεθεί κάποια λύση ώστε να δοθούν τα σωστά κίνητρα. Αντιλαμβάνομαι πόσο ανησυχεί η θα εχουμε καποια προοδο σχετικα συντομα και οτι θα βρεθει καποια λυση ωστε να δωσουν τα σωστα κινητρα αντιλαμβανομαι ποσο ανησυχει η επιτροπη σας στον τομέα αυτών. Συμμερίζομαι τις σας και εύχομαι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το να στηρίζομαι στην ε, παρουσία, στην ε, συζήτηση που θα γίνει στο Συμβούλιο, τίποτε άλλο. Κύριος Κυλακάκης, μίλησε για την ε, πολιτική για το κλίμα που θα χαράξουμε από εδώ και μπρο, στη δεύτερη δηλαδή κλιματική πολιτική και να κοιτάξουμε να στηριχθούμε στι επιτυχίε μα και να διορθώσουμε τα σφαλματά μα. Νομίζω ότι αυτό θέλησα να πω και εγώ στην αρχή τη παρέμβασή μου και συμφωνώ μαζί σα ότι οι αλλαγέ εδώ που αφορούν τις τιμές των βασικών αγαθών και που διαπιστώνονται τα τελευταία χρόνια θα καταστήσει ακόμη πιστεύω πιο ε, αναγκαία την βελτίωση της αποτελεσματικότητας ενέργειας και την αναζήτηση ανάσιμων πηγαίων. Νομίζω επίσης ότι ο στόχος των δύο βαθμών που όλοι πιστεύω επιδιώκουμε σημαίνει ότι κάθε κράτος, κάθε περιφέρεια θα πρέπει να κάνει το μερίδιο της ε, προσπάθειας που της αναλογεί. Αυτό ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για κάθε κράτος, κάθε κράτος έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπισμένο πάντω, ανεξαρτήτως τι κάνουμε με τις ε, πολιτικές για το κλίμα, ότι αυτό θα ήταν προ όφελο τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και αυξήσει μόνο με ρυθμούς αντίστοιχους με αυτούς που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Και ναι, θα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε έτσι ώστε να μην πιέσουμε, να μην συμπιέσουμε μάλλον άλλους τομείς, Φερρυπίν, στο θέμα των υδάτων. Αλλά πιστεύουμε ότι αν δεν τολμήσουμε να επενδύσουμε στο μέλλον τώρα, δεν θα μπορέσουμε να περιμένουμε ε, κάποιες καλές λύσεις, κάποιες ουσιαστικές λύσεις τα επόμενα 10-15 χρόνια. Ελπίζω να απάντησα σε ερωτήσεις όλων σας. Εάν όχι, παρακαλώ μου το θυμίστε. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ακούσουμε τώρα το δεύτερο γύρο. Ο κύριος Καλ Χάντς παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και πάντοτε χαίρομαι όταν μιλάτε για στόχους και αναθεώρηση των στόχων, γιατί με τα προβλήματα που έχουμε δει μέχρι τώρα, ίσως θα ήταν καλό να αλλάξουν κάποια πράγματα. Και βεβαίως υποστηρίζω το προσδιορισμό ρεαλιστικών στόχων στην Ευρώπη για το 2000 ή για οτιδήποτε άλλο. ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε ως Προεδρεύον στο Συμβούλιο και όχι ως Δανός ως προς το θέμα της ε, υλοποίησης των νομοθεσιών ως εθνικό δίκαιο. Αν κοιτάξουμε δηλαδή τι είδους πολιτική για το κλίμα έχουν θεσπίσει τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία, ε, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που έχουν να κάνει και δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα τα μέτρα. Και μπορεί να μιλάμε για 20%, μπορεί να μιλάμε για 30%. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι τίποτε το το θαυματουργό αυτό που βρέθηκε. Και πάντως ε, είναι τόσο ε, υψηλή και τόσο δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι, τόσο δύσκολο να υλοποιηθούν οι στόχοι και δεν χρειάζεται να πάτε μακριά στα καινούρια κράτη-μέλη που βρίσκονται ακόμα μακριά κτλ. Όχι, να πάτε να κοιτάξετε εδώ πέρα, γύρω-γύρω, στο Βέλγιο, στο, στην παλιά Ευρώπη του ΣΥΠΗΝ. Ε, και να δείτε ότι πολλοί απέχουν ακόμη από την ε, προσέγγιση των στόχων. Άρα λοιπόν πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι, συμφωνώ απολύτως. Θα πρέπει όμως και κάποια στιγμή να πούμε ε, από ποιο σημείο αρχίζει το σύστημα λειτουργία, Από πού και πέρα παίρνουμε τα συγκεκριμένα μέτρα και προχωράμε με τα συγκεκριμένα βήματα. Έχουμε ορίσει προστάσει ή καλύτερα διαστήματα πενταετία ή δεκαετία. Έχουμε πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο και θα πρέπει αυτά να τα και χρειάστηκε μάλλον εν τέλει να τα αναβάλουμε, να τα σπρώξουμε μέχρι τέρμα, να τα καθυστερήσουμε όλο περισσότερο και τελικά χρειάστηκε να κάνουμε μια, ένα περιορισμό προς το, στις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα που δεν αδύνατο να τηρηθεί. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι δεν αντιλαμβάνουμε γιατί προσπαθούμε να βρούμε κάτι, πώς μπορούμε μάλλον να βρούμε κάτι που θα ενισχύσει το ETS το οποίο είναι ήδη πολύ αποδυναμωμένο. Μήπως θα πρέπει να βρούμε το θάρρος λοιπόν να πούμε, κοιτάξτε, στον Τέρμαν αποτυγχάνουμε λόγω των ιδιαιτεροτήτων της Πολωνίας. Γιατί διστάζουμε να πούμε ποια είναι η αλήθεια γιατί δεν λέμε ποια είναι ακριβώ η κατάσταση και με ποια βάση μπορούμε να προβούμε σε διαπραγματεύσει. μπορούμε να βγούμε στι διαπραγματεύσει. Εσεί, λοιπόν δεν είστε εδώ ω δανό υπουργό, τουλάχιστον για μένα είσαστε προεδρεύον του Συμβουλίου. Και ω τέτοιο θα ήθελα να μιλήσετε. Και πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υπομονή και την ανοχή σα. Καλώ, λέει ο πρόεδρο, αλλά παρακαλώ τώρα να περιοριστούμε όλοι στα δύο λεπτά για να αφήνουμε του αδελφού να μιλούν. Ο κύριο Γιώργενσον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και για την ε, παρουσίαση. Πολύ χαίρομαι που βρίσκεσαι εδώ στις Βρυξέλλες. Ακούσαμε ότι υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα σε αυτά που θέλουμε σε παγκόσμιο επίπεδο και απ' την άλλη ε, του στόχους τους οποίους πρέπει να πετύχουμε για να ε, μην υπάρχει κλιματική αλλαγή, για να μην προχωρήσει περισσότερο. Υπάρχει η διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για μένα αν δεν πετύχουμε τότε μπορούμε να μιλήσουμε πραγματικά για αποτυχία. Μπορείς να μας πεις λίγο περισσότερο τι θα γίνει με αυτό, τη διαδικασία CCC, τα τρία C. Έπειτα. Πολλέ περιοχέ του κόσμου και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύουν ένα σωρό χρήματα για να επιδοτούν τα στερεά καύσιμα. Μπορεί να μην το ξέρουν πολλοί πολίτε, αλλά είναι τρελό Ορισμένοι μάλιστα ε, δίνουν περισσότερα χρήματα για τα στερεά καύσιμα από ότι για την πράσινη ενέργεια. Ε, αυτό μπορούμε να το ανατρέψουμε και ελπίζω η Προεδρία της Δανίας να το βάλει σε προτεραιότητα στην ημερήσια της διάταξη. Τέλος, είσαι πολύ μετριόφρον και ίσως γι' αυτό να μην το πες στην παρουσίασή σου, εγώ σε γνωρίζω, αλλά θα ήταν χρήσιμο ορισμένοι εδώ να γνωρίζουν τι κάνει η κυβέρνηση στη Δανία. Το λέω γιατί ε, τα ξέρω από μέσα και το πρόγραμμα της κυβέρνησης της Δανίας είναι πολύ φιλόδοξο και πολύ καλό. θα μπορούσες εδώ να το λες. Εντάξει, μην το κάνεις στην Ήτρε, ας πούμε, στη άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά εδώ στη δικιά μας μπορεί να πεις όλα αυτά τα καλά που είναι στο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Κάρλ Σούτερ μετά, αλλά προηγουμένω. ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την εκλογή σα και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Εγώ ήθελα να θέσω μια ερώτηση με κάπω λιγότερο αισιόδοξο από εσά όσον αφορά τα αποτελέσματα του Ντέρμπαν και είμαι πεπισμένο ότι από τη στιγμή που δεν δίνεται μια πολιτική απάντηση στη δήλωση του Μπάλι δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και θα ήθελα κυρίως να Θα ήθελα λοιπόν κυρίως να φτάσω σε μια ουσιαστική απόφαση πιο ισότιμη. Δηλαδή να προχωρήσουμε προς μια απόφαση η οποία θα ληφθεί εν γέννη σύμφωνα με το σύνθημα μιας άδεια εκπομπών για καθέναν ε, και κατά τα λοιπά θα πληρώνουμε. Ε, νομίζω πως κάτι τέτοιο ήταν δίκαιο και ισότιμο για όλους τους πολίτες τώρα εσείς δικαίως θυμήσατε το οδικό χάρτη για το 2050 για μια Ευρώπη άνευ διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση όπου η Διεθνή Συμφωνία φαίνεται να είναι όλο ένα και πιο δύσκολη, γιατί χώρες όπως είπα και ο Καναδάς δεν δέχονται περιορισμούς ε, στην ε, ε, κυριαρχία τους, μήπως θα έπρεπε να αφήσουμε το πρώτο σχέδιό μας για το Κιώτο και να επιστρέψουμε στο δεύτερο σχέδιο, στο πλάνο B, ώστε εμείς να καταφέρουμε για λογαριασμό μας να μειώσουμε και να και όλες ε, τις εκπομπές ε, των αερίων του θερμοκηπίου, να κάνουμε δηλαδή μια πολιτική αυτοπιθαρχίας εδώ στην Ένωση, εσωτερική στην Ένωση και να δώσουμε ε, κάποιες αντισταθμίσεις στις χώρες που δεν δέχονται αυτή την αυτοπιθαρχία όσον αφορά τις εκπομπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το κύριο πρώτη και τώρα ο κύριος Σλιούτερ και μετά η κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ. Δεν είναι θέμα δεξιάς αριστεράς, είναι θέμα ποιος είναι έξυπνος και ποιος όχι. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία στην κρίση που βρισκόμαστε. Τώρα για το πώς θα βρούμε χρήματα. Τα συνταξιδιωτικά ταμεία. Γιατί να μην επενδύσουν στην πράσινη νερή και στο πράσινο μέλλον εφόσον έχουν χάσει τόσα στο χρηματιστήριο. Ίσως να είναι μια καλή επένδυση αυτή. Πάντως, η ιδέα αυτή της πράσινης ανέπτυξης. Ας υποθέσουμε ότι πετύχει, ας υποθέσουμε ότι όλα αυτά τα χρήματα οδηγήσουν στο να πληρωθούν όλα τα χρέη και ότι έχουμε ανάπτυξη 8%. Και μετά πώς θα μειώσουμε κατά 2 με 3% το χρόνο της εκπομπές. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Συνήθως λέμε 1,5-2% ε, αποτελεσματικότητα για κάθε ευρώ. Αν όμως ε, έχουμε τέτοια ανάπτυξη, πώς θα γίνει αυτό. Ένας άλλος τρόπος είναι να αφήσουμε τα πράγματα ε, πιο προσγειωμένα. Ίσως δεν είναι απαραίτητα καλό να αλλάξουμε τα πάντα. Υπάρχουν και όλες αυτές οι νέες πηγές εστερεών καυσίμων. Αν αυτές χρησιμοποιηθούν οι καινούριε, δεν θα καταφέρουμε να μειώσουμε. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε τις ε, σπάνιες γιές, και όλες τις ε, νέες αυτές ε, μορφές που σιγά σιγά έρχονται στο προσκήνιο. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Υπουργός υπογράμμισε την σημασία της ε, πάρκιας ε, ενέργεια και τον, τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, για να εξοικονομηθεί ενέργεια αλλά και οικονομική οικονομικοί πόροι αλλά και για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης που είναι τόσο σημαντικές σε μια, στη σημερινή κατάσταση κρίσης. Συμφωνώ με τη στρατηγική και με τους στόχους και θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι ώστε να να καταφέρουμε να κάνουμε μία ε, εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον της τάξης του 20% μέχρι το 2020. Αλλά επίσης θεωρώ πως είναι απαραίτητο η, τα κράτη-μέλη να ε, προωθήσουν κοινωνικούς στόχους μέσα στο πλαίσιο των μέτρων που προτείνουν για να επιτύχουν τα στόχους της ε, ενεργειακής επάρκειας μέσω συγκεκριμένα της συμπερίληψης μέσων που θα απευθύνονται στους ε, οικογένειες που επηρεάζονται από την έλλειψη ενέργειας και από τις, την ευάλωτη του θέση κοινωνικά. Ποια είναι τα μέτρα και τα συγκεκριμένα κίνητρα που θα δώσετε για τις πιο ευάλωτες ομάδες, ώστε να μπορέσουν δηλαδή να αυξήσουν την ενεργειακή επάρκεια στα σπίτια τους, αλλά και να μειώσετε το κόστος ε, του λογαριασμού της κατανάλωσης ενέργειας. Γι' αυτό το θέμα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάση έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω μία ερώτηση, κάτι σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος ε, Λικάουτ για τις επιδοτήσεις για το πάγο μαγιών. Είπατε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το χάρτη πορείας, μετά την ενεργειακή απόδοση και μετά ε, την αγρανάπαυση. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η αγρανάπαυση πάει για την επόμενη Προεδρία. Θα έλεγα ότι δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα φιλόδοξο αυτό για μια περιβαλλοντική πολιτική, τουλάχιστον όχι τόσο φιλόδοξο όσο θα περίμενα από την Προεδρία της Δανίας. Έχετε κάποιο σχέδιο Β, πλαν B, τι θα κάνετε αν αποτύχει. Έχετε καμιά ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια ευκαιρία στην Ευρώπη να κρατήσουμε τις εκπομπές μας τη δεκαετία αυτή σε τέτοια επίπεδα ώστε να ανταποκρινόμαστε στα όρια του BBC έτσι όπως ε, τα πρότεινε. Ευχαριστούμε κύριε Χάση. Ακουμάτε. Ευχαριστώ λέει η κυρία Μορκουνάιτε. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την ε, ενέργεια, ε, για το πρασίνισμα της Ευρώπης, για την ανταγωνιστική και δυναμική Ευρώπη. Κάτι σε σχέση με τις πράσινες τεχνολογίες. Θέλω να μάθω για την υποδομή ηλεκτρισμού. Αν πρέπει να πάρουμε μαζί αποφάσεις ενία, θα λύσουμε πολλά προβλήματα. Η Δανία θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στις ενεργειακές νησίδες και στη δημιουργία ενός κοινού δικτύου ενέργειας. Νομίζω ότι θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει με μία φωνή με τους προμηθευτές. Ευχαριστώ. Ε, και καλά και κακά νέα. Την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσουμε ε, για το διοξίδιο του άνθρακα στην Επιτροπή αυτή, εφόσον δεν έχουν κλείσει τα πάντα εδώ στο Βέλγιο λόγω της ε, γενικής απεργίας. Ελπίζω να εγκριθεί και στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο ολόκληρο αυτή, αυτός ο χάρτης πορείας. Οπότε η Επιτροπή θα ετοιμάσει τις προτάσεις της για να γίνει πιο αυστηρό το ETS, το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών. Το βέβαια θέμα είναι το Συμβούλιο τι θα κάνει. Θα μπορούσατε εσείς να πείσετε την Πολωνία και άλλους να εγκρίνουν και αυτοί το χάρτη πορείας. Το κακό νέο Μιλούσα με υπαλλήλους από το πρόγραμμα CCST και ζήτησα μια αξιολόγηση για την ανάπτυξη νέων ε, σταθμών ενέργειας υπάρχει μεγάλη ε, αβεβαιότητα. Οπότε δεν ξέρει κανείς να επενδύσει, να μην επενδύσει. Αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα παντού, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χώρες σαν την Πολωνία και όχι μόνο, είναι χώρες για τις οποίες πρέπει να ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον. Δεν πρέπει να είναι ο άνθρακας. Αν όμως τα κράτη-μέλη μπλοκάρουν τις εναλλακτικέ για την ενέργεια, θα έρθουμε αντιμέτωποι πολύ σύντομα με πολύ σοβαρά προβλήματα. Χρειαζόμαστε επενδύσεις και θέλουμε τον χάρτη πορείας για το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Ευχαριστούμε. Τέλος κρίτων Αρσένης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Υπουργό που ήρθε εδώ. Εύχομαι καλή τύχη στις εργασίες σας και για την Προεδρία και για τη Δανία γενικότερα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί. Είναι τα αποτελέσματα του Ντέρμπαν. Φυσικά και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το ότι βρέθηκε στο κέντρο προσοχής η Ευρώπη και για το ότι η στρατηγική ήταν επιτυχής προκειμένου να πετύχουμε συμμαχίες για το χάρτη πορείας. Λέτε και το 2 εφόσον έχουμε χάρτη πορείας. Ε, λοιπόν, εμείς πήραμε το χάρτη πορείας, δεν δώσαμε το και το 2 όμως. Έχουμε μια συμφωνία για μια δεύτερη περίοδο δέσμευσης. Σημειώσαμε τις τροπολογίες που είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας. Το πλαίσιο μένει να αποφασιστεί και έχουμε και την προθεσμία της 1ης ε, Μαΐου για την υποβολή του περιεχομένου. Ποιες θα είναι οι δεσμεύσεις μας για την μείωση των εκπομπών. Συνεπώς, εάν στο Κατάρ τελικά θα βρεθούμε πάλι να μιλάμε με τους συμμάχους μας, θα πρέπει μέχρι την 1η Μαΐου να έχουμε δώσει κι εμείς κάτι σημαντικό. Γι' αυτό ξαναθέτω το ζήτημα το οποίο και εσείς θέσατε εν μέρη. Θα αλλάξουμε κάτι, θα βάλουμε ως προτεραιότητα αυτό το 30% στην ατζέντα ή τέλος πάντων τι θα προσφέρουμε εμείς. Όταν θα έχουμε δηλαδή το χάρτη πορείας θα έχουμε αναλάβει κάποια δέσμευση πριν την 1η Μαΐου για μια δεύτερη περίοδο δέσμευσης. Ευχαριστούμε Κρήτονα. Επιτρέψτε μου να διατυπώσω και εγώ μια ερώτηση. Έχουμε πια την συνθήκη της Λισαβόνας ως υλικό, βαλίτσα με την οποία κυκλοφορούμε. Ίσως μερικές φορές να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει κιόλα. Έχουμε νέα θεσμικά όργανα όπως την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Μπορούμε να υπολογίζουμε στη δική σας στήριξη από την Προεδρία ότι ε, με την διάσκεψη για το κλίμα μπορείτε να αναπτύξετε να, ή να πιέσετε για την ανάπτυξη μιας ε, διπλωματίας για το κλίμα την οποία θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε για ουσιαστικά αποτελέσματα και στη σχέση μας με τρίτα κράτη. Το έχετε αυτό στις ε, προθέσεις της Προεδρίας. Και αν κοιτάξουμε τις ε, προτάσεις της ε, Προεδρίας, το πρόγραμμα της Προεδρίας, έχουμε κλίμα, ενέργεια και κτίρια στις αρμοδιότητές σας, κλίμα, ενέργεια και κατασκευές, που βέβαια έχουν ακριβώς τη θέση τους εδώ. Συγκεκριμένοι στόχοι λοιπόν για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα είναι πράγματα τα οποία έχουμε συστήσει πολλές φορές στο Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι είναι ο κατάλληλος δρόμος και τώρα το σύστημα ανταλλαγής βέβαια, το ETS που συζητήθηκε και νωρίτερα. Όμως, από την κατάσταση του ETS αυτή τη στιγμή και τις δυσκολίες που έχουμε γενικότερα, κινδυνεύουμε από το ενδεχόμενο να πέσει το ETS ε, ε, θύμα της ίδιας της επιτυχίας και να παράγονται ή να ανταλλάσσονται όλο και λιγότερα πιστοποιητικά. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, είμαστε στο 7 ευρώ, Στο 7 ευρώ. Εάν μέχρι το τέλη του χρόνου δεν κάνουμε τίποτα ουσιαστικό, θα περάσει και θα περάσουν και οι θαλάσσιες μεταφορές στο πακέτο αυτό του ETS. Ε, μπορείτε να κάνετε κάποιες προτάσεις για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Παρακαλώ. Κύριος Λίντεγκάρτ. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω ότι είναι 27 χώρες στο Συμβούλιο. Εγώ είμαι μία χώρα. Αν με ακούσετε να σας μιλάω ως Δανός υπουργό, θα πάρετε διαφορετικές απαντήσεις από αυτές που παίρνετε όταν σας μιλάω ως ε, Προεδρία. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό μπορώ να κάνω τώρα, να σας μιλήσω από την ιδιότητα ε, του, της Προεδρίας. Λοιπόν, τι συμβαίνει, τι γίνεται στη χώρα. Θα ξέρετε ότι όταν μιλάμε για τους στόχους του Κιώτο, είμαστε στο δρόμο να ανταποκριθούμε. Το ίδιο και όσον αφορά τους στόχους μας για το 2020 για το διοξίδιο του άνθρακα και για τις ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας. Όχι όμως για την αποτελεσματικότητα. Εδώ ναι, χρειάζεται πρόοδος περισσότερο για την οδηγία αυτή. Κύριε Γιόγκρινσον. Ναι, ε, γνωριζόμαστε από παλιά. Με ρωτάτε, μα τι θα γίνει με το χάσμα αυτό από τώρα μέχρι το 2020, δεν είναι μεγάλη πρόκληση. Ναι, είναι μια μεγάλη πρόκληση, συμφωνώ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε περισσότερα στην Ευρώπη. Και όλοι ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπολογίσει ότι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε μέχρι το 2050 είναι τουλάχιστον να έχουμε 25% μείωση του διοξιδίου του άνθρακα στο εσωτερικό μέχρι το 2020. Αυτό το έχουμε υπολογίσει, το ξέρουμε και αυτό προτείνουμε, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Βέβαια μετά πρέπει να δούμε τι γίνεται και απ' έξω. Στηρίζω όλη τη δουλειά που έχει γίνει προκειμένου να μειωθούν οι επιδοτήσεις για τα στερεά καύσιμα και το στηρίζουμε αυτό. Έχουμε σημειώσει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι και οι Μεξικανοί ακολουθούν την ίδια πορεία ενώπιση του 2020 και ίσως δεσμευτούν και αυτοί σε συνεργασία. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την ε, αεροπλοεία. Υπάρχουν δυνατότητες να καλέψουμε το χάσμα και θέλουμε να το κάνουμε. Ο κύριος Πρόντι με ρωτάει, ο Ιταλός συνάδελφος, τι γίνεται με την ε, διαρροή άνθρακα. Ε, λοιπόν, όλο το σύστημα ETS είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να δεχτούμε την προσέγγιση γιατί ξέρετε ότι δεχόμαστε και την βαριά βιομηχανία και το κάνουμε και στη νέα περίοδο από το 2013 μέχρι το 2020 για την ε, βιομηχανία Έχω ακούσει πάρα πολύ καλές προτάσεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από τη Σουηδία άκουσα κάτι καλό. Πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτήν την μείωση του δεξιού του άνθρακα αν έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση της Δανίας αποφάσισε παρόλο που έχει την ανάπτυξη, να διπλασιάσει τις προσπαθίες της. Τα τελευταία 20 χρόνια βλέπουμε ότι ενώ η βιομηχανία στην αρχή ήταν πολύ επιφυλακτική, σήμερα μας πιέζει να διπλασιάσουμε τους στόχους. Οπότε, εφόσον περάσει το νομοσχέδιο που έχουμε τώρα στη Δανία, θα έχουμε 14% μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και συγχρόνω έχουμε ανάπτυξη. Νομίζω λοιπόν ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Δεν είναι θέμα ανάπτυξη, είναι θέμα τι είδου ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο ανάπτυξη που είχαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά χρειαζόμαστε καινοτομία, ε, ανάπτυξη τη τεχνολογίας και ευημερία είναι μέρος των στόχων μας. Η συζήτηση βέβαια είναι μεγάλη, μπορώ να τη συνεχίσω μαζί σας ε, κάποια άλλη στιγμή. Για την κυρία Στέλλα τώρα. Μιλάτε για την κοινωνική διάσταση όλων αυτών και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά έτσι όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, αν τώρα ε, σταματήσουμε οι τιμές των αγαθών, τροφίμων, ε, ενέργειας κλπ. θα αυξηθούν. Και ο πρώτος που θα πληγεί και θα χάσει έσοδα είναι οι πιο φτωχοί. Αν δεν κάνουμε τίποτα, αυτοί που έχουν να χάσουν περισσότερα είναι οι πιο φτωχοί. Γι' αυτό και πρέπει να επενδύσουμε και να κάνουμε κάτι. Έπειτα πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι πιο ευάλωτοι της κοινωνίας μας θα έχουν τη δυνατότητα και αυτοί να επενδύσουν στην ασφάλεια, την ενεργειακή. Οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν εδώ. Χρειάζεται κατάλληλη κατοικία, Άρα επενδύσεις και επιχειρήσεις που θα βοηθήσουν έτσι ώστε και οι πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού να μπορέσουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους για τη θέρμανση, ηλεκτρισμό κλπ. Συνεχίζω. Α, ναι, η κυρία Χάση. Για την αγρανάπαυση. Και άλλοι με ρωτήσατε για το ETS, το σύστημα ανταλλαγών εκπομπών. Και να πω και για τον κύριο Φλόρενς, ως πρόεδρος του Συμβουλίου, μπορώ βέβαια να διευκολύνω τη συζήτηση, μπορεί να κάνω μια προσπάθεια και θα την κάνω ώστε να προχωρήσουμε γι' αυτό. Και ο καλύτερος τρόπος είναι, και εδώ απαντάω και σε μια άλλη ερώτηση, όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, αυτό το σύστημα έχει δύο στόχου. Ο ένα είναι να διασφαλίσουμε μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αν ήταν αυτό ο μόνο στόχο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχει σημασία ποια είναι η τιμή στην αγορά άνθρακα. Από την άλλη μεριά όμω υπάρχει και ο άλλος στόχος και αυτό είναι να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις ενέργειας και η βιομηχανία στην Ευρώπη θα κάνουν έγκαιρα τι κατάλληλε επενδύσει, ώστε να έχουμε ε, επάρκεια στην, στον εφοδιασμό και κατάλληλες επενδύσεις. Τα επόμενα 20 χρόνια τα δύο τρίτα θα έχει αλλάξει στην Ευρώπη και όσον αφορά την, ε, τον εφοδιασμό ενέργειας. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε φτηνή, καθαρή και ασφαλή ενέργεια. Τέτοιο εφοδιασμό. Αλλιώς ξεχάστε την ανάπτυξη, ξεχάστε την κοινωνική διάσταση ξεχάστε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αλλά βέβαια πρέπει όλοι να συμφωνήσουν στο Συμβούλιο. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να κοιτάξουμε προσεκτικά όλες τις δυνατότητες που έχουμε και να είμαστε ξεκάθαροι για τις συνέπειες της κίνησης που κάναμε είτε για τον άνθρακα, είτε για το EDTP. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρο το τι είναι αναγκαίο. Τι χρειάζεται για να λειτουργήσει το ETS. Εσείς το ρωτήσατε αυτό, Πρόεδρε. Ή όχι. Ποιος το ρώτησε. Α, ο κύριος Ντέιβις, ε, νομίζω τι θα χρειαστεί, πόσος χρόνος θα χρειαστεί. Μα πρέπει να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα πριν πάω στους συναδέλφους στο Συμβούλιο και προσπαθήσω να τους πείσω για το πώς θα προχωρήσουμε. Τι άλλο Επίσης ρωτάτε κατά πόσο ξεγελάσαμε τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Κοιτάξτε, ήμουν και εγώ στις διαπραγματεύσεις με την Προεδρία των χωρών αυτών και ξέρω τι είναι αυτό που τους μοιάζει. Και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι περιμένουν από εμά αποτελέσματα. Δεν νομίζω όμως ότι το κύριο ζήτημα εδώ είναι το αν εμείς θα έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία τους υποσχεθήκαμε. Σίγουρα θέλουν να ακούσουν όμως και τι χρηματοδότηση θα κάνουμε στις δικές τους περιοχές και το τι θα κάνουμε και μετά το 2015. Τι μπορούμε να κάνουμε μαζί με τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες πώς μαζί η Ευρώπη και εκείνη θα μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη ιδίως στις δικές τους χώρες ώστε να μειωθεί εκεί η ένδια που είναι μια από τις προτεραιότητές τους. Και πιστεύω ότι η συμμαχία αυτή θα επεκταθεί περισσότερο και θα αναπτυχθεί περισσότερο. Και ότι αυτό θα γίνει και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Δανίας. Θα φροντίσουμε να φέρουμε σε πέρας τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους συμμάχους μας. Τέλος, Πρόεδρε, ρωτήσατε για την κλιματική διπλωματία. Αυτό που έχω εδώ να σας πω είναι ότι αυτό το οποίο κάνουμε και στο COP17 και αυτό που μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια αυτών των νέων συμμαχιών που αναπτύσσουμε Εννοείται ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το διεθνές πλαίσιο, αλλά σωστά λέτε ότι πρέπει να δούμε αλλιώς και σε άλλα πλαίσια τους συμμάχους μας. Κοινοβούλιο με κοινοβούλιο, κυβέρνηση με κυβέρνηση, έτσι ώστε να υπάρξει οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Όντω. Αυτά νομίζω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σας ε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Λίδεγκαρτ. Σα ευχόμαστε μια πολύ πολύ επιτυχή Προεδρία. Ήταν πολύ επιτυχής η παρουσία σας εδώ. Πολλές και πολυσχηδείς ερωτήσεις διατυπώθηκαν, απαντήσατε με τρόπο πολύ επακριβή, συγκεκριμένο και πλήρη. Και νομίζω μπορούμε και για την ε, πολιτική για το κλίμα και για την ενέργεια όμως να περιμένουμε πολύ καλή συνεργασία με σας. Και όταν υπάρχει μια φιλόδοξη ε, προεδρία για την ενέργεια, για το κλίμα. Είμαστε στο πλευρό σας, μπορείτε να είσαστε βέβαιος ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας είναι στο πλευρό σας. σας ε, ε, εύχομαι λοιπόν κάθε επιταχία, Είναι σαφές ότι η Προεδρία σας είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη για αυτό το εξάμεινο της Προεδρίας και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να βοηθήσετε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η Ευρώπη στα θέματα του κλίματος της ενέργειας ε, και εύχομαι κάθε επιτυχία και συνεργασία με τους συναδέλφους σας από τις άλλες 26 χώρες μέλη. Ευχαριστώ πολύ. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε σε ένα θέμα πολύ συγκεκριμένο και πολύ ε, τυπικό και γι' αυτό πρέπει και το χρόνο να προσέχουμε πάντα, την ακρόαση δηλαδή υποψηφίων εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντο. Έχουμε έξι προσκεκλημένου προσκαλέσει σήμερα. Σα καλωσορίζω όλου. Εδώ. Καθένα από του υποψηφίου έχει στη θέση του 20 λεπτά Αρχίζουμε την ακρόαση με μια πρώτα τρίλεπτη παρουσίαση του κάθε υποψηφίου και στη συνέχεια με τη σειρά μεγέθους ή ομάδες θα διατυπώσουν τις ερωτήσεις τους με τη μορφή του πινκ-πονγκ. Ερωταπόκριση δηλαδή. Και μετά θα πρέπει να ξέρετε ότι 45 λεπτά, δευτερόλεπτα έχετε για την κάθε ερώτηση και ένα λεπτό για την κάθε απάντηση. Είναι πολύ αυστηρά λοιπόν οι συνθήκες, οι όροι για την ακρόαση αυτή. Παρακαλώ να τηρηθούν. Παρακαλώ λοιπόν οι ομάδες να φροντίσουν να είναι εδώ παρόντες όσοι έχουν δηλώσει πως θα καταθέσουν ερώτηση και τον πρώτο υποψήφιο μπορούμε να τον ακούσουμε τώρα, πρόκειται για τον κύριο Ρινάλτο Ζενούγουα, ο οποίος έχει το λόγο για μια παρουσίαση τρίλεπτη για να ακούσουμε στη συνέχεια τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Ρινάλτο Ζενεβουά και διδάσκω μηχανική γεωλογία στο τμήμα γεωφύλου φυσικής στο, στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα της Ιταλίας. Βρίσκομαι εδώ ως ε, υποψήφιο ε, αντιπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Ε, για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί αυτός ο οργανισμός μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ηγετικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος καθώς και ε, της ε, ανθρωπότητος. Ε, η μελλοντική μου εργασία, εάν εγκρίνεται αυτή την υποψηφιότητά μου, είναι να εξασφαλίσω ότι ο αέρας, η γη και το νερό, για να συνοψίσω, θα αποτελούν αντικείμενο προσοχής για όλους μας, έτσι ώστε οι αυρινές ε, γενναίες να κληρονομήσουν ένα καθαρότερο και γέστερο κόσμο. Ωστόσο, ε, η αναπόφευκτη υπόσχεση βιώσιμης ανάπτυξης δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς συντονισμένες και συγκεκριμένες προσπάθειες για τη μετόπιση των ε, περιβαλλοντικών πολιτικών για την γνώση και κατανόηση της φύσης ε, στην ευρεία της έννοιας και των ανθρωπογενών επιπτώσεων στην ίδια τη φύση. Αυτές οι επιπτώσεις είναι περίπλοκες ε, και δύσκολο να προβλεφθούν ε, λόγω του μεγάλου αριθμού μεταβλητών και αγνώστων παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση. Απορρέει λοιπόν η ανάγκη για συλλογή πληροφοριών, στοιχείων που θα πρέπει να οργανωθούν κατά τέτοιο τρόπο και να ερμηνευθούν από εμπειρογνώμονες ώστε αυτά τα αποτελέσματα να μπορέσουν να γνωστοποιηθούν σε όλους ε, και κατά αυτόν τον τρόπο να εξυπηρετήσουν καλύτερα το διάφορους περιβαλλοντικούς, κυβερνητικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ένα τρόπο για να διαχειριστούμε τη την, ολική, την οικολογική αλληλεπίδραση είναι νομίζω κατάλληλη για αυτό το έργο εάν δούμε το τι έχει γίνει μέχρι στιγμή και το τι θα πρέπει να γίνει προβλέπω μια πολύ δεσμευτική θέση για τα επόμενα τρία χρόνια. Είμαι βέβαιος πω η μακρά μου εμπειρία στι γεωμορφολογικές μελέτε, καθώς και στι υδρολογικές μελέτες και έρευνε, θα με βοηθήσουν σε αυτή την εργασία καθώς επίσης και ο συντονισμός ε, σε διάφορα διεθνή θέματα και συγκεκριμένες μελέτες όπως ε, η σχέση μεταξύ κατολιστήσεων και κλιματικών αλλαγών ή πλημμυρό, η πρόβλεψη πλημμυρών μέσω ε, ειδικών δικτύων. Επίσης για να επιτύχουμε μια πλήρη αμφίδρομη επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα να ζητήσω πάντοτε στην περίπτωση που εγκρίνεται την υποψηφιότητά μου να έχω μια ειδική επαφή, ιδιαίτερη επαφή με τα μέλη του Κοινοβουλίου για άμεσο διάλογο και επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζωνοφό. Και τώρα εκ μέρους των ομάδων. Κύριε Γκαρδίνη πρώτη, από το ΕΛΚ, 45 λεπτά. Δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Eh, σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να αναπτύξετε λίγο περισσότερο γιατί είδα το βιογραφικό σα που είναι εξαίρετο από την ακαδημαϊκή άποψη. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν ποια είναι η συγκεκριμένη σα εμπειρία, η πρακτική σα εμπειρία στα περιβαλλοντικά ζητήματα και θα ήθελα επίση να γνωρίζω πώ θα μπορούσατε να ε, διαρθρώσετε τη σχέση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά κυρίως με εμά, με το Ευρωκοινοβούλιο, για να μπορέσετε να μας ε, καλύψετε τις απαιτήσει των βουλευτών στο πλαίσιο του, της πιο τεχνικής εργασίας που είναι η εργασία του οργανισμού. Η Λίντα Μακάβαν. Μετά. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ακαδημαϊκός, ε, οπότε στην ουσία η κατάρτισή μου αφορά την έρευνα και τις μελέτες. Αλλά όπως συχνά συμβαίνει στην Ιταλία, όλοι έχουμε επαφές με τις περιφέρειες, με την κεντρική κωδικητικό μηχανισμό του Ιταλικού κράτους και γι' αυτό έχω αναπτύξει ιδιαίτερα στον τομέα των κατολιστήσεων και των πλημμυρών, φλάτζ, συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία μπορούν άμεσα να εφαρμοστούν από τις περιφερειακές αρχές και από τις τοπικές αρχές και πιο συγκεκριμένα έχουμε αναπτύξει κάποια προγράμματα παρακολούθησης των, των επιφανειακών κατολιστήσεων υψηλού κινδύνου τόσο λόγω ε, ταχύτητας όσο και λόγω του, του μεγέθους της και παράδειγμα την μελέτη της κατολίσθησης του Βαγιώτη. Εγώ θα ήθελα μέσα στο πλαίσιο αυτής της, του οργανισμού θα ήθελα να έχω πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για το πώς να αναπτύξουμε ε, σχέσεις ανάμεσα σε μένα και στο Κοινοβούλιο και γι' αυτό και ζήτησα συγκεκριμένα την ε, επιλογή ενός προβουλευτή ε, με τον οποίο να μπορώ να συζητήσω ποιες είναι οι ανάγκες του Κοινοβουλίου και ποιες είναι οι επιθυμίες του οργανισμού περιβάλλοντος. Από αυτούς ε, νομίζω πως είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να πω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ζενεβά. Η ε, Λίντα Μακάβαν. Εδώ ε, είμαι. Αριστερά σας. Δεν ξέρω τι επαφές είχατε με τον οργανισμό μέχρι τώρα, αλλά πώς αξιολογείτε το έργο του οργανισμού αυτού. Και αν πάτε εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει κάποια βελτίωση όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού αυτού. Ευχαριστούμε. Απάντηση. Είναι η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με τον οργανισμό. Δηλαδή δεν... και με τούτο το κοινοβούλιο εξάλλου. Κρίνω πως η δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα ο οργανισμός είναι πολύ καλή. Είναι πολύ σημαντική δουλειά που αφορά κατ' ουσίαν ε, τις πτυχές της πληροφοριών και στοιχείων και ε, ερμηνείας εξήγησης αυτών των στοιχείων καθώς και διάδοση ε, των αποτελεσμάτων ε, στα μεμονωμένα κράτη, στο ίδιο το Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν πολιτικές για βιώσιμη ανάπτυξη. Η δουλειά λοιπόν αυτή είναι εξαίρετη. Πώς θα μπορούσα εγώ να βελτιώσω τη δουλειά του οργανισμού. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα φιλόδοξο. Νομίζω πως αυτά όλα θα πρέπει να τα συζητήσουμε συλλογικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και να βρίσκουμε σε στιγμή ποιο είναι η καλύτερη λύση στο κάθε πρόβλημα. Να πω πιο συγκεκριμένα ότι κάτι που θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο είναι να βρεθεί να βρεθούν και να συγκεντρωθούν στοιχεία για ορισμένες πτυχές ε, των επιπτώσεων ε, των ε, κλιματικών αλλαγών για τις επιφανειακές, όπως σας είπα, κατολιστήσεις και πλημμύρες. Μέχρι στιγμής είναι περιορισμένα τα στοιχεία, ακριβώς επειδή πρόκειται για φαινόμενα που είναι πολύ δύσκολα στην ερμηνεία τους. Και ε, στην ε, χαρτογράφησή τους και γι' αυτό, ε, σε αυτό σίγουρα θα ήθελα να προχωρήσει αυτή η δουλειά, να βρεθεί δηλαδή μια ευρωπαϊκή κοινή πολιτική. Και τώρα παρακαλώ την φιλελεύθερη ερώτηση με τον κύριο Γκεμπράντη. 45 δεύτερα η ερώτηση, ένα λεπτό η απάντηση. Χωρίς Παρακαλώ παρατάσεις για να έχουμε την της ευκαιρίες για όλους τους υποψηφίους. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η... πρώτη ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι αυτή που έκανε η Λίντα Μακάβιν, αλλά την απαντήσατε. Η δεύτερη είναι εξή. Πέρα από το επιστημονικό υπόβαθρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν και κάποια ελάχιστη εμπειρία όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους πολιτικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει ο καθηγητής Ζενεβουά, τι εμπειρία έχει στον ευρωπαϊκό χώρο. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, ακούμε την απάντηση. Κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σας και είναι μια ερώτηση πολύ κέρια. Όπως είπα, ήδη. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ από αυτή την ιδιότητα. Είχα άλλες ευκαιρίες να βρεθώ εδώ όταν συντόνισα κάποια προγράμματα ευρωπαϊκής έρευνας για, λόγω των οποίων είχα επαφές αλλά όχι άμεσα με το Ευρωκοινοβούλιο. Από όσο γνωρίζω για τη δομή του Ευρωκοινοβουλίου και για τις σχέσεις ανάμεσα στον οργανισμό και το Κοινοβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και το Κοινοβούλιο προκύπτουν αποκλειστικά από τη δική μου μελέτη στα διάφορα site στο δίκτυο για την ίδια την, τον ίδιο τον οργανισμό και για το κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους των τώρα. Κυρία Χάση. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, από το βιογραφικό σας βλέπω ότι είσαστε ειδικό στη γεωλογία. Αλλά δεν αναφέρονται άλλοι τομείς που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Θα ήθελα λοιπόν να μου κατονομάσετε τρεις μεγάλες προκλήσεις, περιβαλλοντικές προκλήσεις που βλέπετε εσείς και αν έχετε κάποιες ιδέες για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ενημέρωση από τον οργανισμό αυτό προς τους ε, και τους πολιτικούς που παίρνουν τις αποφάσεις αλλά και στο κοινό, προς το κοινό. Απάντηση παρακαλώ. Δεν κατάλαβα καλά. Δεν κατάλαβα καλά την μετάφραση. Εγώ είμαι γεωλόγος. Δεν είμαι τοπογράφος. Προκλήσεις ε, οι κύριες για μένα είναι αυτές που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Όπως σας είπα, τις, που αφορούν κυρίως τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που είναι δύο πτυχές που σχετίζονται, δύο φαινόμενα που σχετίζονται άμεσα με τις κλιματικές αλλαγές. Άλλη πρόκληση είναι είναι η σύλληψη, η συλλογή του διοξιδίου του άνθρακα, όπου η γεωλογία πάλι ε, επεμβαίνει για την αποθήκευση του αερίου αυτού. Και η τρίτη πρόκληση είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι μη ανανεώσιμες. Αυτές είναι πολύ σημαντικές προκλήσεις. Όλες οι προκλήσεις ωστόσο είναι το ίδιο σημαντικές εγώ απλώς ανέφερα αυτές που, για τη δική μου ειδίκευση έχουν ε, μεγαλύτερη σχέση. Η Σιέρα από ό,τι βλέπω δεν έχουν εκπροσώπηση. Ούτε η Γκουε. Ούτε η Εύτη. Και άρα περνάμε στους στους και πάλι Λίντα Μακέιουαν. 45 δευτερόλεπτα. Όχι. Ελκ. Γκαρντίνη. Ε, eh, Εγώ θα ήθελα να επανέλθω λίγο, αν και είπατε ότι δεν έχετε συγκεκριμένη εμπειρία για από αυτόν τον οργανισμό και άρα στις σχέσεις με το Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα. Ωστόσο πιστεύω ότι επειδή αναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους, θα ήθελα να σας ξανακάνω το πρώτο μου ερώτημα, στο δεύτερο του σκέλος. Πιστεύω πως είναι σημαντικό στις σχέσεις με τους οργαν, διάφορους οργανισμούς να έχουμε να συνειδητοποιήσουμε μάλλον πόσο σημαντικός είναι ένας, ε, μια μόνιμη σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο. Διότι έτσι έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και πιστεύω πως αυτό είναι κάτι που το θέλουμε όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο. Γιατί ο οργανισμό σας όχι μόνο θα πρέπει να μας δώσει μέσα για να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε, αλλά και να παρακολουθήσει την κατάσταση στις χώρες για να δει αν και πώς αυτές οι νομοθεσίες εφαρμόζονται και πώς συγκεκριμενοποιούνται τα προγράμματά μας. Κύριε Ζενεβουά, παρακαλώ. Ναι, κατάλαβα καλά την θέση σας αυτή. Η θέση είναι και η δική μου όταν εξέφρασα την επιθυμία να έχω έναν εκπρόσωπο συγκεκριμένο του Κοινοβουλίου με τον οποίο να ενημερώνω και να έχω επαφέ που σίγουρα θα πρέπει να είναι συνεχής και πλήρης χωρίς και χωρίς βέβαια να ξεχνάμε και τη πιθανότητα συμμετοχής ε, πιο συγκεκριμένης και εις βάθος συμμετοχής στην ε, σύνταξη των εκθέσεων ε, του οργανισμού που θα είναι η βάση των γνώσεων που θα έχουμε συλλέξει και που φυσικά θα μπορούν να διανεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες και τους ενδιαφερόμενους για τα αποτελέσματα των μελετών του οργανισμού. Κύριε Ζουνεβά, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ, για την παρουσία παρουσίαση, για τις απαντήσεις. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο υποψήφιο, τον κύριο Χένεκε. Κύριε Πέτερ Χένεκε, παρακαλώ να έρθετε εδώ μπροστά. Η διαδικασία θα είναι ακριβώς ίδια με αυτή που ακολουθήσαμε για τον κύριο Ζουνεβουά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ και που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για αυτήν την τόσο σημαντική θέση εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συνοψίσω καταρχήν κάποια στοιχεία κλειδί όσον αφορά την καριέρα μου. Μετά τον Βάιτσικερ, πρόεδρο του Ινστιτούτου του 2000, ήμουνα πρόεδρος το 2003 μέχρι το 2008 του Ινστιτούτου. Στη συνέχεια άφησα ως εμερίτου στο Πανεπιστήμιο και τώρα δουλεύω σε διάφορα θέματα με για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ατζέντα ακριβώ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Βούπερταλ. με, ασχολούμαι με την εφαρμοσμένη έρευνα όσον αφορά το περιβάλλον. Έχω δουλέψει υπό τον Γιώσκαρ Φίσερ ως εμπειρογνώμων για θέματα ενεργειακής πολιτικής ή και στο τμήμα στρατηγικού σχεδιασμού. Συμμετείχα και σε διάφορα συμβουλευτικά όργανα για εθνικά και διεθνή ε, σώματα. Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, για το κλίμα και την ε, ενέργεια. Και ήμουν μέλος του GF-STEP. Σήμερα δουλεύω ως ε, επιστήμον για θέματα τα οποία έχουν ε, άμεση σχέση με ε, τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Το ένα θέμα είναι η προστασία των πόρων όπου είμαι επικεφαλής ενός ε, μεγάλου προγράμματος γερμανικής εταιρείας που δουλεύει για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επίσης δουλεύω και πάνω στα οικονομικά μοντέλα και τις στρατηγικές επικοινωνίες πάντα για την επάρκεια πόρων στη Γερμανία. Και συμμετέχω και σε ένα μεγάλο πρόγραμμα που ονομάζεται Bridging the Information έχει να κάνει με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Έχει ξεκινήσει από το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος από το 2009 και προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της γνώσης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων σε διεθνές επίπεδο. Και συνεργαζόμαστε με πολλά διεθνή δίκτυα, το SPN, το ESPI και άλλα. Κύριος στόχος μας είναι ακριβώς να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει σήμερα όσον αφορά την κατασκευή κτηρίων σε διεθνές επίπεδο. Άρα είμαστε με πλατφόρμα ε, πληροφοριών που προσφέρει ενημέρωση όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την ε, κατανάλωση, το κόστος, ε, την, την εξοικονόμηση που μπορεί να γίνει κλπ δουλεύουμε και σε συνεργασία και με την Κίνα, την Ινδία και τις Βρυξέλλες βέβαια. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν προσπαθώ να αναπτύξω πολιτικές ενεργειακής απόδοσης και να συνεισφέρω όσο γίνεται περισσότερο στη, στο New Green Deal. Τόσο στη χώρα μου όσο και ευρύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Την και τώρα περνάμε σε ερωτήσεις των ομάδων. Κύριε Γκαρντίνη. Γκουαρντινή για 45 δευτερόλεπτα. Ε, ε, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, προηγούμενο, να ρωτήσω αυτό που ρώτησε και τον προηγούμενο υποψήφιο, γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς το άνθρωπος που θα πάει να δουλέψει στον οργανισμό σκοπεύει να αυξήσει τη δυνατότητα εργασίας και συνεργασίας με το κοινοβούλιο. Ε, ενδιαφέρει λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα από το βιογραφικό σας είδα ότι έχετε, συνεργάζεστε με τον Περιφερειακό Υπουργό. Ε, πώς πιστεύετε ότι μπορούν να εναρμονιστούν οι διαφορές που υπάρχουν ε, και είναι τόσο μεγάλες και ευρείες ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. Είναι πολύ έντονες και προφανείς οι διαφορές και δημιουργούν προβλήματα όταν ε, πρέπει να νομοθετήσουμε για τις 27 χώρες. Ευχαριστώ να ακούσουμε την απάντηση. Χωρίς μικρόφωνο. Ναι, Εάν μιλάμε λοιπόν για την έρευνα, πάντα αυτό σημαίνει, θα ήθελα να αναφέρω, ότι έχω συμμετάσχει και σε ακροάσει ε, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και άλλων διεθνών οργανισμών για να μπορέσω να αποκομίσω το δυνατόν περισσότερη ε, ενημέρωση από την επικαιρότητα, από τον πραγματικό κόσμο του ΣΥΠΗΝ δική μας η πραγματογνωμοσύνη στον Ινστιτούτο του Βούπερταλ ήταν πάντα προσανατολισμένη στην ε, πραγματικότητα, την πολιτική δηλαδή. Ε, πάντοτε κοιτούσαμε να έχουμε απαντήσεις για ερωτήματα που θα ενδιέφεραν ένα κοινοβούλιο, ένα πολιτικό φορέα. Οι διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών είναι τεράστιες, όμως αποτελούν ταυτόχρονα και ένα μεγάλο πεδίο γνώσης για το λεγόμενο leapfrogging, ε, δηλαδή το άλμα του βατράχου. Μεγάλες διαφορές παραγωγικότητας μεταξύ του ε, ασθενέστερου και του ισχυρότερου παραγωγικά κράτους μέλους, 1 προς 9, ακόμα και 1 προς 17. Άρα μπορούμε να διδαχθούμε, πιστεύω, από την εμπειρία των πιο προηγμένων κρατών για το τι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε στην σταδιακή εισαγωγή μιας βιώσιμης ανάπτυξης σε λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη. Ευχαριστώ πολύ. Λίντα Μακέδων. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για την παρουσίαση, για τη δουλειά σας στην πολιτική. Είχατε κάποια επαφή με την υπηρεσία περιβάλλοντος. Και βέβαια η άλλη ερώτηση, όπως και στον προηγούμενο υποψήφιο, τι θα θέλατε να αλλάξει στην υπηρεσία, τι είδους αλλαγές θα επιφέρατε εσείς. Απάντηση. Επαφές με την υπηρεσία περιβάλλοντος ήταν ουσιαστικά επιστημονικού χαρακτήρα. Έχουμε και ε, αποστείλει δικό μας προσωπικό, δικούς μας συνεργάτες στην υπηρεσία περιβάλλοντος Είχαμε πάρα πολύ καλή ε, συνεργασία είτε για σενάρια είτε για δείκτες με βάση αυτά τα οποία έχουμε εμείς ε, διαπιστώσει από την έρευνα στο Βουτπέρθαλ. Άρα είμαστε κομμάτι αυτού του δικτύου που έχει αναπτύξει η υπηρεσία. Και αντίστοιχα έχουμε και το συνδετικό κρίκο με την ε, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία και με την, ε, μεταξύ Ομοσπονδιακής Γερμανικής Υπηρεσίας και υπηρεσίας, ε, αποκεντρωμένης υπηρεσίας της ε, Αυτό που χρειαζεύω είναι μια υπηρεσία περιβάλλοντος η οποία ένας οργανισμός περιβαλλον ο οποίος θέλει σε θέση να συζητήσει ένα νέο Green Deal, ένα νέο σύμφωνο για την οικολογία με δείκτες, με απασχολήση, με αηφορία, πολιτικές αποφάσεις, δηλαδή με βάση και οικονομικούς όρους, χωρίς ε, να μπορώ βέβαια να το χαρακτηρίσω ως αδυναμία μέχρι τώρα της ε, υπηρεσίας, νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί ε, η θεώρηση των οικονομικών παραγόντων. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των φιλελευθέρων κ. Κεμπράντη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον καθηγητή και για τις δηλώσεις του μέχρι τώρα. Έχετε πολύ καλές επιδόσεις πρέπει να πω. Η δική μου ερώτηση αφορά το ρόλο που θα μπορούσατε να διαδραματίσετε στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, ως προς τον προσδορισμό προτεραιοτήτων και για την ε, ίδια την υπηρεσία, για τον ίδιο τον οργανισμό περιβάλλοντος. πιστεύετε ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να θεωρηθεί ότι έχει κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει ο οργανισμός ή θεωρείτε ότι θα έπρεπε σε ορισμένα πράγματα να κάνει κι άλλα, να προχωρήσει ακόμη περισσότερο ή πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχει πολύ πιο σαφή πολιτική, πολιτικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Δεν μπορώ εγώ να αποτολμήσω κάποια διαπίστωση, κάποια κριτική για το αν έχουν σωστά διατεθεί η λίγη, η λιγοστή πόρη που διαθέτει ο οργανισμός. Πάντως, θα έλεγα ότι Εάν κοιτάξουμε τα τρία βασικά σενάρια, δηλαδή ενέργεια, κλίμα και αποτελεσματικότητα στη χρήση των, ε, του, της ύλη των πόρων, ίσως δεν είναι ακόμη ικανοποιητικά τα αποτελεσματά ως προς τους ε, επιδιωκόμενους στόχους αποτελεσματικότητας της χρήσης ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων. Υπάρχουν σενάρια σημαντικά με ιδιαίτερες πολιτικές για τον κάθε τομέα, φερρυπίν, στα ε, κτίρια, φερρυπίν στην διεθνή συνεργασία, διαχείριση γνώσεως όπως λέγεται ή μεταφορά γνώσεως για πράγματα στα οποία η Ευρώπη έχει καλή ε, εμπειρία και μπορεί να την εξαγάγει σε άλλα κράτη λιγότερο προηγμένα. Αυτά, πιστεύω, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ακόμη και οικονομικούς πόρους για τον οργανισμό. Δεν τα έχει όμως ακόμη καταφέρει. Ευχαριστώ πολύ, Σαν το Μάνση. Η κυρία Χάση, συγγνώμη για τους πράσινους. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που βλέπετε και πώς μπορείτε να βελτιώσετε τις ε, πληροφορίες, την ενημέρωση και για αυτούς που είναι υπεύθυνοι να λαμβάνουν αποφάσεις βεβαίως, αλλά και για ε, το κοινό, για τους πολίτες. Απάντηση. Έχουμε να λύσουμε ένα γενικό, ένα κεντρικό πρόβλημα στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ποσοστό ε, προόδου, η, ο λόγος προόδου αύξησης δηλαδή της ε, χρήσης ε, ύλης αλλά και της ε, τη αποτελεσματικότητας μάλλον στη χρήση ενέργειας πρέπει να, είναι, πρέπει να είναι αρνητικός ε, πάντα για να μπορούμε να περιμένουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Από την άλλη, για να δημιουργηθούν νέες εργασία, θα πρέπει να προχωρήσει η παραγωγικότητα της εργασίας χαμηλότερα από την οικονομική παραγωγικότητα. Και άρα η βιωσιμότητα σε κάθε διάσταση, δεν πρόκειται για οικολογική, για οικονομική, για κοινωνική, πρέπει να αντιμετωπιστούν με πραγματική σοβαρότητα και να υλοποιηθούν με σοβαρότητα. Αυτό είναι η κύρια πρόκληση κατά μένα για το περιβάλλον και για την οικονομική πολιτική στη Γερμανία. Πρέπει αυτό το οποίο μπορούμε να περιγράψουμε ως πακέτα κινήτρων, να, και που έχουμε εισαγάγει, θεσπίσει λόγω της κρίσης, να το εμπλουτίσουμε έτσι ώστε να ε, ενισχυθεί το ποσοστό των επενδύσεων, να ξεκινήσει μια πιο δυναμική ή να ταθεί σε κίνηση μια πιο δυναμική διαδικασία που θα οδηγήσει και σε νέες της Ευχαριστώ. Η ακόμη δεν έχουμε, ούτε την ΚΟΕ, ούτε την ΙΕΦΤΗ. Σοσιαλδημοκράτες. Και πάλι κυρία Λίντα Μακέιβεν. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω το βιογραφικό σας. Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου, διαχείρισης, συγκρούς συμφερόντων και άλλα τέτοια διοικητικά είναι τα θέματα που απασχολούν το Διοικητικό Συμβούλιο ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού, όχι επιστημονικά θέματα. Τι έχετε να πείτε λοιπόν. Να σας πω, δεν υπάρχει πιο ε, συγκρουόμενη η, περισσότερη εσωτερική σύγκρουση, περισσότερες εσωτερικές συγκρούσεις ε, υπηρεσία από ό,τι αντίστοιχη γερμανική. Έχουμε πάντα να επιλύουμε στήματα συγκρούσεων. Φερρυπίν το ζήτημα του πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, να προωθήσουμε μια αποτελεσματική πολιτική ενέργειας και πάντοτε καλούμεθα να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Εάν αυτή η Διαρευνητική Επιτροπή την οποία ανέλαβα ε, δεν είχε μπορέσει να σταθμίσει ζητήματα και να καταλήξει σε συμβασμούς δεν θα είχαμε ούτε τη μεταλλαγή στον χώρο της ενέργειας, ούτε θα είχαμε λάβει τις αποφάσεις για την εγκατάλειψη πυρηνικής, ούτε θα είχαμε συνένεση για ε, πολιτική για τους νέους πόρους, για τους ανανεώσιμους πόρους ενέργειας, όπως έχουμε τώρα, όπως έχουμε συμβάλει στο Ρίο ε, 20, που πιστεύω ότι θα μπορέσει ιδιαίτερα να συμβάλλει η ε, Γερμανία και για τους συμβασμούς, αλλά και ιδιαίτερα για τη δυνατότητα που έχει να ε, σταθμίζει καλά διαφορετικά συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον θεωρώ πως ήταν το έργο της ζωής μου και έχω πολύ μεγάλη εμπειρία από την αντίστοιχη επιτροπή, από τις αντίστοιχες επιτροφές, επιτροπές ε, πραγματογνώμων, όπως ονομάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Γκουαρντίνη, όχι, δεν έχετε ερώτηση. Συμπληρωματική ερώτηση έχετε. Όχι, καλά είμαι, ευχαριστώ. Καλώς ευχαριστώ. Κλείνει ο γύρος των ερωτήσεων και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Χένικε για τις ερωτήσεις, την παρουσίαση. Ας δούμε τώρα τον τρίτο. Υποψήφιο Κρίστιαν Χάι. Sie Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να σας ε, παρουσιαστώ για αυτή την πολύ σημαντική θέση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Καταρχήν ε, να σας πω ότι είμαι Γενικός Γραμματέας του Γερμανικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου για το Περιβάλλον που είναι για την Γερμανία, στην Γερμανία ένα ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο το οποίο ορίζει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και για να αξιολογεί την κατάσταση του περιβάλλοντος για να προειδοποιεί την κυβέρνηση και το ευρύτερο κοινό για τις ε, εξελίξεις και για να δίνει συστάσεις για πολιτική. Η σημερινή μου εργασία αφορά το συντονισμό 7 πανεπιστημιακών καθηγητών από, διάφορες εργασίες, από διάφορους τομείς, ε, φυσικές επιστήμες, ζωολογία κτλ. και να καθοδηγώ την δουλειά αυτών των επιστημόνων. Η συμβουλευτική μου εργασία ανήκει μέσα στο, μάλλον συνεργαζόμαστε διαρκώς με το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, διαρκώς χρησιμοποιούμε τις εκθέσεις του και τις εφαρμόζουμε στο εθνικό ε, πλαίσιο. Τα τελευταία δέκα χρόνια επίσης έχω, έχω διατελέσει σε ηγετικέ ε, θέσεις σε Ευρωπαϊκά Συμβούλια για το Περιβάλλον, που είναι ένα δίκτυο τέτοιων συμβουλίων ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή προεδρεύω του ομάδα Εργασίας για την Ενέργεια σε αυτό το δίκτυο. Εργαζόμαστε για τις βιώσιμες υποδομές για την Ευρώπη, καθώς επίσης για την οικονομία, για τον οδικό χάρτη για την οικονομία χαμηλού άνθρακα μέχρι το 2050. Ως Ευρωπαϊκό Δίκτυο έχουμε τακτικές επαφές με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και έτσι είμαι αρκετά εξοικειωμένος με την εργασία του οργανισμού αυτού. Προσωπικά Είμαι επιστήμων ειδικευμένος στις ευρωπαϊκές, στην ανάλυση ευρωπαϊκών ε, πολιτικών περιβάλλοντος και θέματα ε, διακυβέρνησης στην επιστημονική μου εργασία τα τελευταία 20 χρόνια έχω καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ε, περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και μεταφορών και ενέργειας από την ευρωπαϊκή οπτική. Από το 1997 μέχρι το 2001 ήμουν ε, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ομοσπονδιακού ε, Περιβαλλοντικού Γραφείου είχα εντατικέ επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και έχω την αίσθηση ότι έχω μια κάποια συνέστηση και κατανόηση των αναγκών και των προοπτικών των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού ε, Οργανισμού Περιβάλλοντος. Εμένα μου αρέσει πολύ η συνεργασία με αυτόν τον οργανισμό γιατί πιστεύω πως κάνει εξαίρετη εργασία και γι' αυτό και ενδιαφέρομαι για αυτή τη θέση. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να στηρίξω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει τις ανάγκες του μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορώ να επενδύσω χρόνο και ενέργεια για να το κάνω αυτό και έτσι νομίζω μπορώ να βοηθήσω το Ευρωπαϊκό Οργανισμό να καταστεί ισχυρότερος και να είναι ένας σημαντικός ε, παίκτη μέσα στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ε, πάνω απ' όλα πιστεύω πως η πρόκληση είναι το θέμα της άβλησης των επιπτώσεων των αλλαγών του κλίματος. Έπειτα έχουμε τη συζήτηση για την πράσινη οικονομία και θα ήθελα να αναφέρω και ένα τρίτο θέμα που για μένα σημαντικό. Πρόκειται για την ολοκληρωμένη εποπτεία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Και περνάμε στο γύρο των ερωτήσεων και πάλι Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κύριε Κουαρτίνη. Σα Σας ευχαριστώ. Δεδομένης της μακράς σας ήθελα να σας ρωτήσω πώς πιστεύετε πως θα μπορούσατε να βελτιώσετε την, το έργο αυτού του οργανισμού να φτάνει δηλαδή περισσότερο σε εμά που πρέπει να νομοθετήσουμε, αλλά και στους πολίτες που συμμετέχουν ε, άμεσα, γιατί οι περιβαλλοντικές πολιτικές τους επηρεάζουν άμεσα. Δηλαδή, ποια θα μπορεί να είναι η δική σας προστεθέμενη αξία, αν ε, ε, μπαίνατε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ευχαριστώ πολύ. Επάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος κάνει κατα... πάρα πολύ καλό έργο, εξαιρετικό έργο, περίπλοκο πεδίο πολυσχηδείς πληροφορίες και δεδομένα επεξεργάζεται και από αυτά προκύπτουν και τα πολιτικά μηνύματα. Αυτά θα αποστολούσαν για μένα μια βάση κίνησης. Έχω την αίσθηση πάντως ότι τα δεδομένα αυτά δεν φτάνουν μέχρι την κοινή γνώμη όπως θα έπρεπε ε, και δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ο οργανισμός περιβάλλοντος θα αναλάβει και το έργο αυτό μόνος του. Θα πρέπει με την επαφή με τις εθνικές υπηρεσίες και τα focal points, τα σημεία εστίασης, να επικεντρωθεί στην έκφραση του μηνύματος, ε, των μηνυμάτων αυτών κατά τρόπο ουσιαστικό και κατανοητό για την κάθε χώρα, για την κοινή γνώμη της κάθε χώρας. Αυτό θα ήταν μια από τις προτεραιότητες κατά με. Επίσης βλέπω στο πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά καιρού να δίνεται έμφαση στον τομέα των ε, υπηρεσιών οικοσυστημάτων της πράσινης οικονομίας. Είναι σαφής το μήνυμα ότι δηλαδή εξαρτάται η οικονομία μας από τα παρθένα οικοσυστήματα. Ταυτόχρονα όμως πέραν αυτής της δήλωσης με το σαφής ε, και τη συζήτηση για την πράσινη οικονομία θα πρέπει να δώσουμε και πιο πολύ ουσία ε, και εμπειρική ε, και με εμπειρικό τρόπο ε, να εμπλουτίσουμε τις ε, υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε για τα οικοσυστήματα. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών και Ελληντά Μακέβαν. Σαφώς έχουμε μεγάλη εμπειρία, έχετε μεγάλη εμπειρία στην Ευρωπαϊ... για τα ευρωπαϊκά θέματα και γνωρίζετε τον οργανισμό πολύ καλά, οπότε δεν θα ρωτήσω το ίδιο που ρώτησα τους υπόλοιπους υποψηφίους. Ε, είδατε ότι στα θέματα περιβάλλοντο έχουμε κάνει κάποια πρόοδο στην Ένωση, αλλά κοιτάζοντα προ το μέλλον, ποια θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στο μέλλον. Τα πάει καλά η Ένωση στο περιβάλλον. Μπορεί να κάνει περισσότερα. Πώ βλέπετε να προχωρούν τα πράγματα. Αν έγινε πρόοδο στο παρελθόν θα μπορέσουμε να κάνουμε παρόμοια πρόοδο και στο μέλλον, νομίζετε. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν είναι τόσο απλό, διότι τα απλά προβλήματα Μπορεί να τα έχουμε λύσει απλά προβλήματα, είναι αυτά τα οποία μπορεί κανείς να επιλύσει με τεχνικού χαρακτήρα μέτρα. Αυτά που έχουμε μπροστά μας όμως τώρα είναι τα πολύ πιο δύσκολα, τα λεγόμενα έμμονα προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή αξιοαπορίας ότι η οδηγία για τη χρήση των γεών δεν έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, ότι δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα τα σχετικά με την προστασία των οικοσυστημάτων, την ε, μη υπερβολική αποψήλωση των δασών. Όλα αυτά είναι τομείς δηλαδή πολύ πιο δύσκολοι και γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη δουλειά στην διαμεσολάβηση και στην ενημέρωση, στην επικοινωνία δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους των φιλελευθέρων. Γκεμπράντι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ για τη μέχρι τώρα παρουσίασή σας. Έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά τον σημερινό σας ρόλο στο Γερμανικό Συμβουλευτικό ε, Συμβούλιο μάλλον ε, για το περιβάλλον. Αυτό το Συμβούλιο είναι εξάρτητο από την κυβέρνηση και το ρωτώ έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων στο μέλλον και ε, έπειτα βλέπω την εφαρμογή την, ως μία από την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής ε, Νομοθεσίας. Εσείς βλέπετε ότι θα είχε κάποιο ρόλο να παίξει ο Οργανισμός Περιβάλλοντος όσον αφορά την καλύτερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στην Ευρώπη. Συμβουλή μου είναι και αυτό νομίζω το λέξε καθαρά η οδηγία είναι ότι θα πρέπει να επικρίνουμε μια κυβέρνηση. Το πράγμα άλλωστε και τακτικά. Είχαμε παραδείγματι μια έκτακτη ε, έκθεση που δημοσιεύτηκε λίγο πριν από την Φουκουσίμα και που επέκρινε την στάση προς τα πυρηνικά της ε, κυβέρνησης. Είμαστε με ένα διοικητικό τμήμα του, ε, του κράτους, δηλαδή της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, αλλά δεν έχουμε υποταγή από την διοικητική υπαγωγή. Είμαστε ανεξάρτητοι δηλαδή. Τώρα, εάν θα πρέπει ο οργανισμός περιβάλλοντος να δίνει κρίσεις, να εκδίδει κρίσεις για το που σημειώνονται πρόοδος και που όχι, πιστεύω ότι είναι ότι μπορώ να είμαι σύμφωνος, αλλά χρειάζεται και περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές που βλέπονται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και πλέον η ιδέα της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και ενός τέτοιου οργανισμού θα κινδύνευε αν ε, παρενέβαινε υπερβολικά στον έλεγχο της εκτέλεσης ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το θέμα της εκτέλεσης, της επαλήθευσης εκτέλεσης ε, εμπίπτει σε αρμοδιότητες κάποιου άλλου ευρωπαϊκού οργάνου. Ευχαριστώ για τους πράσινους κυρία Χάση. Ευχαριστώ. Θέλω να ακούσω και από εσά, παρακαλώ, Πώς ε, βλέπετε εσείς τρεις σημαντικές προκλήσεις για το περιβάλλον και πώς πιστεύετε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα μπορούσε να βελτιώσει την ενημέρωση για αυτά τα θέματα και την επικοινωνία μαζί μας που παίρνουμε τις πολιτικές αποφάσεις αλλά και με το κοινό. Με την συζήτηση για το κλίμα, αν κοιτάξουμε έναν ορίζοντα μέχρι το 2005, έχουμε πιστεύω μπροστά μας ουσιαστική ανάπλαση, αναδιόρθωση των υποδομών μας, του τρόπου ζωής και αυτό αποτελεί έργο Ηράκλειο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ταυτόχρονα δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα δημιουργώντας πρόβλημα κάπου αλλού. Η κλιματική αλλαγή δηλαδή πάντοτε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ταυτόχρονο μέλημα για την διαφύλαξη της βιοποικιλότητας. Γιατί αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα του πώς μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα δημιουργώντας ένα άλλο πρόβλημα όπως φερειπίν στα γεωργικά καύσιμα, βιοκαύσιμα και άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης μεγάλη πρόκληση είναι ο ρόλος της Ευρώπης ως προς την υπέρβαση αυτού που ονομάζουν οι επιστήμονες ασφαλή πλανητικό, ασφαλές πλανητικό όριο. Υπάρχει ένα σημείο καμπής από το οποίο και μετά μπορεί να χαθούν πάρα πολλά για την ανθρωπότητα. Μεγάλο πρόβλημα θα είναι παραδείγματι και το άζωτο και το διοξίδιο του θείου και άλλα αντίστοιχα προβλήματα, αλλά και η χρήση των γεών. Ευχαριστώ. Η CR δεν έχει. Η FD όχι. Κουε όχι. Και προχωρώ. Κυρία Μακέιβον. Όχι. Δεν έχετε ερώτηση. Γκαρντένι. Όχι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν κύριε για την παρουσίαση, για τις απαντήσεις σας. Τέταρτος υποψήφιος τώρα. Κύριος Χολτσπικ. Καθίστε, πάρτε μια ανάσα και ξεκινάμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ονομάζομαι του Χόσπετ, Ο κύριος ε, τομέας ε, πραγματογνωμοσύνης μου είναι τοξικολογία του περιβάλλοντος. Τελευταία μάλιστα τα έχετε συζητήσει κι εσείς αυτά. Επίσης είμαι οικολόγος που ε, δουλεύω και εργάζομαι όσον αφορά τις νυχτερίδες και τα δελφίνια και ασχολούμαι με τα είδη των οικοτόπων που έχουν να κάνουν με την οδηγία για τους οικοτόπους και για την ε, βιοπικιλότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκίνησα τη συνεργασία μου με την Επιτροπή σας πρώτα απ' όλα όταν είχαμε την οδηγία REACH και τις ρυθμίσεις για την προστασία από τα παρασιτοκτόνα. Είχαμε 1.400 προτάσεις για να αλλάξει το REACH. Θυμόσαστε ότι ήταν δύσκολη η διαδικασία. Χάρη όμως στην Επιτροπή αυτή πετύχαμε καλά αποτελέσματα. Βέβαια, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια πράγματα όπως είναι ε, τα ε, νανοσωματίδια, ε, οι φαρμακευτικές ουσίες που ακόμα θέλουν ε, δουλειά. Σίγουρα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στήριξης της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον. Ο κύριος στόχος πάντως των ε, εκπροσώπων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, είναι ακριβώς ο οργανισμός να κάνει αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί να κάνει. Να μην ε, αποκτήσει μια δικιά του ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να εκφράσω κάποιες ανησυχίες για το τελευταίο πρόγραμμα εργασίας όσον αφορά το 2012. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος σίγουρα είναι από τους καλύτερους. Σίγουρα έχει πολύ καλό κόσμο που δουλεύει εκεί, καλή επιστημονική γνώση και αποτελέσματα, αλλά, αλλά πρέπει να υπάρχει και ρεαλισμός δεδομένου ότι ξέρουμε ότι ο προπολογισμό δεν θα αυξηθεί. Άρα ο οργανισμός πρέπει να δρά με σοφροσύνη στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την σύντομη και λεπτομερή σας εισαγωγή. Θα αρχίσουμε τώρα το γύρο των ερωτήσεων. Η κυρία Καρδίνη πρώτα, εκ μέρους του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξέρω πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε την συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ. Πώς ε, θα υπάρξει δηλαδή περισσότερη διαφάνεια, καλύτερη σύνδεση και ανταλλαγές απόψεων. Γιατί αν δεν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, χάνονται μεγάλες ευκαιρίες. Απάντηση παρακαλώ. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτιωση. Πιστεύω ότι η δουλειά που γίνεται είναι τέλεια η επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο γιατί όλους μας εξυπηρετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί ακόμα. Αυτό όμως που κυρίως μπορεί να βελτιωθεί είναι ο οργανισμός να μας προσφέρει περισσότερα σενάρια. Την πολιτική δεν την αποφασίζει ο οργανισμός, εσείς ε, την αποφασίζετε την πολιτική. Συνεπώς θα μπορούσε να ενισχυθεί ε, το ίχνος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος εδώ. Υπάρχει πάντα ένας σύνδεσμος, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες συναντήσεις με προσωπικό από τον οργανισμό, ανάμεσα δηλαδή στον οργανισμό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, ίσως θα μπορούσε η γραμματεία σας να έχει την επαφή αυτή. Πάντως εκεί θα μπορούσε να υπάρχει πραγματικά βελτίωση στο θέμα της επαφής. Ευχαριστούμε. Η Λίντα Μακέβεν εκ μέρους των Εσείς δεν ξέρω πόσο συχνά ε, πρέπει να πηγαίνετε στο Διοικητικό Συμβούλιο, πάντως αυτό που είναι ενδιαφέρον αυτό που είπατε, ότι δηλαδή πρέπει να παραμείνει στο δρόμο του Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και ότι είναι επικίνδυνο γιατί μερικές φορές ε, παίρνουν το δικό τους δρόμο ανεξάρτητα από αυτό για το οποίο έχουν φτιαχτεί, γίνονται περισσότερο αυτόνομοι. Εσείς πιστεύετε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό. Πιστεύετε δηλαδή ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα το κάνει αυτό για τον οργανισμό. Εγώ είχα πάει ως αντικαταστάτης όντως και είχαμε αποφασίσει ο Μιχάλης Κούρος ήταν εκείνος που ήταν πάντα περίπου στις συναντήσεις παρακολουθούσα και εγώ το Επιστημονικό Συμβούλιο και αντικαταστούσα όταν κάποιοι δεν μπορούσαν να πάνε. Πήγα, όχι στο 100%, αλλά στις περισσότερες από τις συναντήσεις για τις οποίες είχα προβλεφθεί, οι περισσότερες ήταν όντως του Επιστημονικού Συμβουλίου. Και συγχρόνως με αυτό που έκανε ο Μιχάλης, και εμείς μπορούσαμε έτσι να καταλάβουμε πολύ καλά τι έκανε ο οργανισμός. Και η ανησυχία μου ήταν, α, επευκαιρία να σας πω πρώτα απ' όλα, ότι ήταν εξαιρετικό το έργο, αλλά εδώ δεν θέλω να είμαστε σε μια εικονική πραγματικότητα. Σημαντικό είναι η επικοινωνία μας με το κοινό. Οι αναφορές online στην ιστοσελίδα είναι κάτι πάρα πολύ καλό, δεν λέω, αλλά κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να υπάρχει πραγματική επαφή. Με τις περικοπές Πρέπει κανείς βέβαια να επικεντρώνεται στον κύριο ρόλο του. Έχετε την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ναι, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνετε το κύριο σας καθήκον, να αναλάβετε την πρώτη σας αρμοδιότητα και να τη φέρετε σε πέρες. Εκ μέρους των φιλελεύθερων τώρα, ο κύριος Γεμπραντή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ κύριε Χόλσμπεκ για την παρουσίασή σας. Έχουμε συνεργαστεί τα τελευταία δυόμιση χρόνια πολύ με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζω ήδη κάποιες από τις ε, ιδέες σας αυτά τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Έχω όμως μία ερώτηση για τις προτεραιότητες μέσα στον οργανισμό. Πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να αλλάξουν? Μιλήσατε για την επαφή με το κοινό και για τον ψηφιακό τρόπο επαφής είχατε κάποια επικριτική σε αυτό. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος ρόλος όσον αφορά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ότι δηλαδή ο οργανισμός έχει κάποιο ρόλο στην ε, θέση σε ισχύ της νομοθεσίας. Απάντηση. Ο προϋπολογισμός θα σταθεροποιηθεί στα επίπεδα του 2011, μια πολύ μικρή αύξηση, όχι ουσιαστική, για την υπηρεσία στην Κοπεχάγη βέβαια. Αυτό είναι κρίμα γιατί έχουν αρμοδιότητες και για τις κλιματικές αλλαγές. Συνεπώς, με αυτές τις ευθύνες και αρμοδιότητες ε, των εκθέσεων που πρέπει να ετοιμάζουν, πρέπει να υπάρξει ε, κάποια ιεράρχηση. Θα πάνε στην πάντα κάποιες ε, δράσεις, θα μπουν σε προτεραιότητα κάποιες άλλες. Έτσι κι αλλιώς πρέπει τα αποτελέσματα να είναι υψηλής ποιότητας. Μερικές φορές όταν κανείς προσπαθεί να ικανοποιήσει πολλούς και να κάνει πολλά πράγματα, πέφτει ποιότητα. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος. Ευχαριστούμε για τους πρασίνους τώρα. Η κυρία Σατοχάση παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Είπατε ότι ο οργανισμός πρέπει να ιεραρχήσει τις αρμοδιότητες της. Μπορείτε να επεκταθείτε περισσότερο. Τι εννοείτε με αυτό. Είπατε επίσης ότι τις επαφής online, ε, την επαφή αυτή, τις εκθέσεις online, δεν είναι κάτι που για σας θα είναι προτεραιότητα. Πώς μπορεί να βελτιωθεί πάντως η πληροφόρηση από πλευρά του οργανισμού προς τους πολιτικούς και προς το κοινό. Τα επιστημονικά ζητήματα πώς θα γίνει να είναι πιο σαφή. ώστε να τα αντιλαμβανόμαστε καλύτερα. Απάντηση. Συμφωνώ ότι η επικοινωνία με το κοινό είναι πάρα πολύ σημαντική και για τον οργανισμό. Συνεπώς, φυσικά και πρέπει το μήνυμά σας να περάσει με στοιχεία τα οποία να στέκουν επιστημονικά. Πρέπει να είσαστε και προσεκτικοί για το τι θέλετε να κάνετε. Για παράδειγμα το θέμα ε, του θορύβου. Εγώ ευχαρίστως να συμμετέχει και το κοινό και με τα κινητά Το ένα θέμα το οποίο προέκυψε από το Κοινοβούλιο και στη συνέχεια ήταν υποχρέωση του οργανισμού να πει στο Κοινοβούλιο ότι δεν υπήρχε επιστημονική βάση για να γίνει κάτι τέτοιο τη συγκεκριμένη στιγμή. Συνεπώς, πρέπει να ιεραρχήσει κανείς τις προτεραιότητές του. Ποιες είναι πώς μπορεί να συνεισφέρει επίσης σε σενάρια έτσι ώστε να σας παρουσιάσει εσά τα διαφορετικά σενάρια και τη σχέση κόστους και ωφέλους, χωρίς βέβαια να πληγεί η οικονομία. Και όταν έχετε τα σενάρια, εσείς οι πολιτικοί θα αποφασίσετε από εκεί και πέρα τι θα κάνετε. Εκεί βλέπω εγώ να έχει αρμοδιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε. Από την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά. Δεν βλέπω κανέναν. Και άρα έχει δυνατότητα οι σοσιαλδημοκράτε να θέσουν άλλη ερώτηση. Όχι. Κύριε Γκουαρδίνη, επίση θέλει. Σα ευχαριστώ θερμά. Κύριε Χολσπίκ, για τη συμμετοχή σα εδώ, για τι απαντήσει σα και για το ότι τηρήσατε το χρόνο Πέμπτος υποψήφιος, παρακαλώ. Κύριος Σκόλος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βέβαια ότι είστε κουρασμένοι. Θα προσπαθήσω όμως να επαναλάβω μερικά από αυτά τα οποία ήδη έχω σημειώσει στο βιογραφικό μου και να επικεντρωθώ στο γιατί κάνω αίτηση και πάλι. Είμαι χημικός, περιβαλλοντολόγος χημικός και ωκεανογράφος με ιδιαίτερες, ε, ιδιαίτερη εξειδίκευση στο θέμα του περιβάλλοντος και ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση. Ε, είμαι καθηγητής του Πανεπιστήμιου των Αθηνών, διδάσκω περιβάλλον και ωκεανογραφία η UNESCO μου πρότεινε πρόσφατα μια έδρα διαχείρισης για βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης και επίσης ε, ιδιαίτερα συμμετέχω και σε οργανώσεις, συνεργάζομαι και με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με τα θέματα αυτά. Πολλά είναι τα χρόνια στα οποία αφοσιώθηκα στην εργασία σε διάφορες οργανώσεις όπως το Ευρωπαϊκό ε, Γραφείο Περιβάλλοντος που ανέφερε και ο Κρίστιαν και έχω την μοναδική και μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ το σώμα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος από την πρώτη συνεδρίασή του. Ένας από τους λόγους για τους οποίους επανέρχομαι ως υποψήφιος είναι ότι Πιστεύω πως έτυχα της εμπιστοσύνης του, της Επιτροπή Επιτροπής των Προέδρων από την πρώτη εποχή με τον Κεν Collins και τον Καρολάιν Jackson μέχρι το Γιολάινεν. Και επίσης, διότι πιστεύω βάσιμα πιστεύω ότι έχω συμβάλει στην ανάπτυξη και την ε, διαμόρφωση από πλευρά σας αυτού του οργανισμού που είναι πιστεύω ακράδαντα επιτυχής και ότι πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Θα ήθελα επίσης να πω ότι αποφάσισα να επαναθέσω υποψηφιότητα, γιατί είναι πολύ δυσχερή ο ρόλο, πιστεύω, να σα εκπροσωπεί κανεί στο κοινό, στο, στον οργανισμό και θα εξηγήσω γιατί. Και πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχεια στο έργο αυτό. Πρόκειται για έναν οργανισμό αρκετά περίπλοκο. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή μέσα σε δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στον χρόνο συν άλλες δύο του εκτελεστικού Προεδρείου να αντιληφθεί το περίπλοκο χαρακτήρα και τις δομές ε, του οργανισμού, άρα χρειάζεται κανείς περισσότερο χρόνο και έτσι χρειάζεται, εάν αποφασίσετε να ε, με ορίσετε και πάλι ως εκπρόσωπό σας, να προβλέψετε μια δυνατότητα αλλά ε, μέσα σε, με, μέσω των προσώπων, δύο τακτικών, δύο αναπληρωματικών, αλλά πάνω απ' όλα και χρόνο, τρεις εβδομάδες το χρόνο ή περισσότερο, επαρκεί για την επικοινωνία. Διότι πρέπει και εσείς να συμβάλλετε ουσιαστικά, όχι απλώς να έχετε μία παρουσία, αλλά να είστε παρόντες, να διαβάζει κανείς τις εκθέσεις, να ε, κάνει σχόλια, να ε, έχει την επικοινωνία με όσους από εσάς εδώ στο Κοινοβούλιο ενδιαφέρεστε πράγματι. Και καθώς είχαμε τον κύριο Γκερμπράντι ως υποψηφίο, ως εκπρόσωπό σας, νομίζω ότι ήταν πολύ καλή αυτή η δυνατότητα. Πρόεδρε, τελειώνω. Τέσσερα λεπτά είχατε πει. Τρία λεπτά. Μάλιστα, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ορίζεται κάποιος υποψήφιος, αυτό προβλέπει ο υποψήφιος εκπρόσωπος, ε, αυτό λέει ο τίτλος ε, της ακρόασης, αλλά ουσιαστικά είμαστε οι η ψυχή σας εκεί, η παρουσία σας εκεί πρέπει να καταλαβαίνει κανείς και τα δύο όργανα, και τον οργανισμό και το κοινοβούλιο και να μπορεί να εξασφαλίζει και την ε, ισορροπία μεταξύ και της εκπροσώπησης της Επιτροπής και του, των συμφερόντων ή του συμφερόντος των κρατών μελών, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σταματώ λοιπόν εδώ. Ασφαλώς θα έχετε και εσείς πολλές ερωτήσεις. Ίσως μπορέσω να επεκταθώ περισσότερο στα άλλα θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάθε υποψήφιος έχει μόνο τρία λεπτά. Και θέλω να είμαστε όσο δυνατόν. Να έχουμε ισότητα μεταχείριση για τον καθένα. Καλώς. Και τώρα περνάμε στο γύρο των ερωτήσεων. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει το λόγο πρώτα με την κυρία Γκουαρτίνη. Ναι, σας ευχαριστώ. Κατάλαβα ότι εάν ε, συνεχίσετε στο Διοικητικό Συμβούλιο θα μας δώσετε πολλές ε, πληροφορίες. Φαντάζομαι πως οι στάσεις θα είναι τα ίδια και όσον αφορά τι, που κατά πόσο θα εισακούγονται τα όσα σας λέμε εδώ, γιατί θα πρέπει να τα μεταφέρετε σε αυτόν τον οργανισμό. Πέρα από τις ε, ικανότητές σας, ποια είναι άλλη τομή ενδιαφέροντο σας και να κάνω και την ερώτηση που έκανα και στον προηγούμενο υποψήφιο. Κατά τη γνώμη σας, καθώς είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει στο έπακρο τους πόρους που έχει στη διάθεσή του, ποιες θα ήταν οι προτεραιότητες που θα μας δίνατε εσείς. Παρακαλώ να απαντήσετε σε ένα λεπτό, κύριε Σκούλο. Όπως είπα ήδη, έχω καλύψει πολλούς τομείς πέραν των υδάτων στο έργο μου. Όλες τις πτυχές του περιβάλλοντος, πολλή δουλειά στα μέταλλα, ήμουν και στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για την ε, τοξικότητα και οικοτοξικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολλά άλλα όργανα και φορείς διαχειριστικούς ή άλλους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχει σημασία το δεύτερο κομμάτι της δεύτερης σας, ε, το δεύτερο κομμάτι της δηλαδή προτεραιότητες. η ιδιαιτερότητα είναι ότι δεν μπορεί κανείς να περιορίσει ένα κομμάτι. Πρέπει να επεκτείνει το έργο του σε όλους τους τομείς, δηλαδή και περιβαλλοντικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες απαιτούν να προσφέρει πληροφορίες στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, αλλά και λόγω των προτεραιοτήτων των κρατών. Δηλαδή είμαστε μέσω του ορισμένο από εσάς εκπροσώπου και, της, ε, και του Προεδρείου της Επιτροπής ή του Προέδρου της Επιτροπής σε επικοινωνία με το Κοινοβούλιο για να ακούμε τις δικές σας προτεραιότητες και να τις μεταφέρουμε στο έργο της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μακέβαν, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Έχετε πολλά χρόνια εμπειρία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τι έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει προτεραιότητες. Τι προτεραιότητες πρέπει να έχουμε για το μέλλον, κατά την άποψή σας. μεγάλη αλλαγή. Καταρχάς, μπορώ να σας πω ότι ένα από τα κύρια μελήματα ήταν το κοινοβούλιο να είναι το όντι παρόν και να εισακούγεται ε, ισότιμα με τους άλλους και την Επιτροπή. Μου ζητήσατε να μιλήσω, να, θέσω το ζήτημα της υλοποίησης, δηλαδή ενός τύπου monitoring, παρακολούθηση των ε, πολιτικών που δεν ήταν δυνατόν στην αρχή. Μπορέσαμε να τα καταφέρουμε. για τα σενάρια ε, αλλά και με διάφορους τρόπους ε, παρακολούθησης που όμως ε, φτάνουν και μέχρι την ε, διεθνή, τις διεθνείς σχέσεις, τη διεθνή εικόνα του περιβάλλοντος, δηλαδή τη λεγόμενη περιβαλλοντική διπλωματία. Αυτή είναι νέη τομείς και πρέπει να προχωρήσουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ε, ευκαιρίες που έχουμε, νέες τεχνολογίες και ισορροπία νέες τεχνολογίες αλλά και γνώση, διάδοση της γνώσης αυτής στο ευρύτερο κοινό. κοινό. Ο κύριος Γκερμπάντη έχει το λόγο των φιλελευθέρων. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Σκουτό για όλη τη δουλειά που έχει κάνει τόσα χρόνια Πραγματικά δραστηριοποιηθήκατε στον οργανισμό και κάνατε πολύ καλή δουλειά. Δεν έχω ερωτήσεις να σας κάνω γιατί έχουμε συνεργαστεί στενά τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Ίσως ε, για τους συναδέλφους να ρωτήσω το εξή. Έχετε την αίσθηση πως ο οργανισμός μπορεί να γίνει ακόμα ισχυρότερος ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να περιοριστεί στον ρόλο που έχει σήμερα. εγώ νομίζω πως μπορεί να καταστεί ισχυρότερος χωρίς να ξεπεράσει το ρόλο του όπως αυτός περιγράφεται στον καρονισμό. Μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός. Ως οργανισμός χρειάζεται να είμαστε περισσότερο παρόντες στις πρωτεύουσε με την έννοια ότι κάποια από τη δουλειά που κάνουμε δεν χρησιμοποιείται και αυτό είναι ευθύνη τελικά των διαφόρων πρωτευουσών, των κρατών μελών. Αλλά και εμείς ως οργανισμός μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω μέσω διαφόρων ε, καναλιών. Επίσης πρέπει να προσεγγίσουμε άλλους ενδιαφερόμενους ε, εφορείς με πιο δραστήριο τρόπο και αυτά όλα μπορούν να γίνουν μέσα στο πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο που ισχύει ήδη και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε τον οργανισμό. Και επίσης γνωρίζετε πολύ καλά πως υπάρχουν ορισμένοι τομείς όπου χρειάζεται να περιοριστούμε ώστε να ενισχύσουμε κάποιους τομείς όπου χρειάζεται καινοτόμως εργασία. Ένα από τα βασικά προβλήματα, όχι προβλήματα μάλλον, προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο οργανισμός είναι ότι χρειάζεται να είμαστε γενικά στην ε, πρωτοπορία. Γιατί είναι ένα τομέα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο και αυτό πρέπει πάντοτε να το έχουμε υπόψη μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πράσινη. Κύριε Χάση. Ευχαριστώ. Καθηγητά Σκουλέ, θα ήθελα να σας ακούσω επειδή ήσασταν ήδη αρκετά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερό σας επίτευγμα κατά τη διάρκεια αυτών των ετών στον οργανισμό. Χωρίς μικρόφωνο, ο κύριος Κουρλός. Σας ευχαριστώ. Ειλικρινά, αν επισκεφθείτε τον οργανισμό θα δείτε ότι οι απόψεις του Κοινοβουλίου εισακούγονται. Και τολμώ να πω ότι εισακούγονται επί ίσης ώρες με την γνώμη της Κομισιόν και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα έχουμε σχηματίσει μια κουλτούρα συνεργασίας και συνένεσης και νομίζω πως αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα όσον αφορά τη δική μου συμβολή, αν αυτό είναι που με ρωτήσατε τώρα. Ποια είναι τα επιτεύγματα του οργανισμού εν γέννη. Είναι πολλά. Το πρώτο είναι ότι έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες, που τώρα δεν είναι απλά πληροφορίες, αλλά κινούνται προς την σωστή ερμηνεία και μια ολόκληρη σειρά, όχι όλες, αλλά μια ολόκληρη σειρά χρήσιμων σενάριων ε, για τη λήψη αποφάσεων ε, και ταυτόχρονα καταφέραμε να δώσουμε χρόνο για επιπλέον αιτήματα από το Κοινοβούλιο μέσα στο πλαίσιο του ετησίου προγράμματος εργασίας. Υπάρχει δηλαδή πάντοτε ε, χώρος για νέα μελέτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακόμη δεν έχουμε κανέναν από τους η EFD, του CCR και την ΚΟΕ και γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα για άλλη μια φορά από τους Ολυδημοκράτες την κυρία Ελίνα Μακέβαν. Έχετε καμιά ερώτηση. Όχι, ούτε η κυρία Κουαρτίνη από ό,τι βλέπω. Και ως εκ τούτου σας ευχαριστώ θερμά κύριε Σκουλό για την παρουσίαση, για την απάντηση σε ερωτήσεις σας. Και περνάμε στον έκτο ψήφιο, κύριο Πιέρ Βέλιγκερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, αγαπητοί Ευρωβουλευτές. Υπομονετικά θα πρέπει να με ακούσετε. Για να σας πω τα Πρώτα απ' όλα, η δέσμευσή μου για το περιβάλλον είναι μεγάλη. Γι' αυτό και θέλω να δουλέψω εκ μέρου σα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Γιατί, γιατί είμαι τόσο υπέρ του περιβάλλοντος. Σε τρία επίπεδα συμβαίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα, εκεί που ζω, ζω σε ένα χωριό στι κάτω χώρε στην Ήπεθρο, εκεί προστατεύω το, το περιβάλλον και το τοπίο, αλλά και ως πολίτης Είμαι ενεργός πολίτης σε διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τόσο στη χώρα μου όσο και διεθνής. Και συνεργάζομαι με άλλους επιστήμονες και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την ε, ολοκληρωμένη αξιολόγηση στο κέντρο Τίντελ, για παράδειγμα. Με τον Ρίκο Ματέπιση στην Ιταλία, όπως το ΕΚΟ στη Γερμανία. Και έχουμε αναπτύξει μια μέθοδο πώς δηλαδή να συμπεριλάβουμε περισσότερο τα περιβαλλοντικά ε, ζητήματα στην Ευρώπη. Από το 1997 μέχρι το 2005 και είχαμε αυτή την μέθοδο και τώρα ακόμα και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος την χρησιμοποιεί. Επίσης θέλω έναν ισχυρό ρόλο του Κοινοβουλίου για το Περιβάλλον. Να υπάρξει εναρμόνιση μεταξύ των χωρών, αλλά και σε διεθνέ επίπεδο, Ντέρμπαν και άλλες διεθνείς συμβάσεις υπέρ του περιβάλλοντος. Ο Ευρωπαϊκός Αυτός Οργανισμός Περιβάλλοντος αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για να βελτιώσουμε την ποιότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα της λήψης αποφάσεων για θέματα περιβάλλοντος. Θα είναι τιμή για μένα να σας εκπροσωπεί εκεί. Και δεσμεύομαι να έρχομαι εδώ θα έρχομαι. Ξέρω ότι έχετε, εσείς δεν προλαβαίνετε δεν μπορείτε να έρχεστε. Εγώ θα έρχομαι αρκετές φορές μέσα στον χρόνο και θα συζητάω μαζί σας και θα φροντίσω να υποστηρίξω τις απόψεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον οργανισμό. Λοιπόν, σας είπα ότι είναι προσωπική μου πεποίθηση. Δεύτερον, πιστεύω στην Ευρώπη και την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και τρίτον θέλω τη δικιά μου γνώση και εμπειρία να την χρησιμοποιήσω και να την προσφέρω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τελευταία δύο χρόνια έχω κερδίσει πολλή εμπειρία ε, σε θέματα περιβάλλοντος μέσω της επιστήμης. Για 20 χρόνια παρακολουθώ το έργο του οργανισμού από την αρχή. Καταρχήν ήμουν διευθυντής στο τμήμα περιβάλλοντος των κάτω χωρών. Και θυμάμαι ότι τότε είχαμε συζητήσεις για το πού θα γινόταν αυτός ο οργανισμός. Ήταν ή η Βαρκελόνη ή η ε, Κοπεχάγη. Μετά κάτι ήταν και για τη Βουδαπέστη. Στη συνέχεια αργότερα ε, επιστήμων, αλλά και τώρα είμαι επικεφαλής ενός Εθνικού Προγράμματος Έρευνας για το κλίμα στις κάτω χώρες. Με 100 εκατομμύρια. Και συνεργαζόμαστε και σε διεθνές επίπεδο, με το ΕΚΟ, με το ΤΙΛ και άλλα Ινστιτούτα, στην Πολωνία, στην Ισπανία και αλλού. Στις κάτω χώρες Δουλεύω με διάφορα τμήματα και οικονομικών και υδάτων και μεταφορών. Ε, συμβουλεύω για την πολιτική τους και για θέματα επίσης ρήπανσης του αέρος ή μόλυνσης των υδάτων. Τέλος, τέλος, ελπίζω να μπορέσω να σας εκπροσωπήσω και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε και αρχίζουμε τις ερωτήσεις. Πρώτον, η κυρία Κουαρδίνη, εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι λίγο δύσκολο τώρα να κάνουμε ερωτήσεις σε αυτή τη φάση. Ήδη απαντήσατε σε πολλά από τα πράγματα που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ωστόσο, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε καλύτερα την ε, σχέση ανάμεσα εφόσον είστε καδημαϊκός και μελετητής, πώς βλέπετε την, ε, την εφαρμογή όλων αυτών ε, στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Γιατί ανάμεσα στις ΜΚΟ, ε, ε, τον ακαδημαϊκό κόσμο και τους πολιτικούς ε, φαίνεται να μπερδεύονται τα πράγματα όσον αφορά τη συγκεκριμενοποίηση των προγραμμάτων. Δεν ξέρω αν σας εκφράστηκα αρκετά καλά με καταλάβετε. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι βομβαρδίζεστε από προτάσεις και από πληροφορίες Οπότε εδώ ακριβώς είναι που ο οργανισμός περιβάλλοντος μπορεί να ε, διοχετεύσει καλύτερα τις πληροφορίες αυτές και σε συνεργασία με τα Εθνικά Ινστιτούτα. Έχω δει πώς δουλεύουν και πώς ε, έχουν ε, βελτιωθεί, αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν υπάρχει επαφή με εθνικούς βουλευτές και με εθνικέ οργανώσεις. Πρέπει το έργο να είναι αποτελεσματικό και για σας και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει μια γενική συνένεση με τα εθνικά Ινστιτούτα για το ότι είναι σημαντικό και τι είναι δευτερεύον. Γι' αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός μπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο σε αυτό και να ξεχωρίσει την ύρα από το στάρι. Δηλαδή εκείνες τις προτάσεις που είναι πιο ενδιαφέρουσες από εκείνες που είναι λιγότερο. Ευχαριστούμε. Εκπέρους των Σοσιαλιστών τώρα, Λίδα Μακάβιν. Στη χώρα σας δραστηριοποιήσετε πάρα πολύ για το περιβάλλον. Πιστεύετε ότι το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο, πιστεύετε ότι είναι κάτι που εσείς θα χρησιμοποιούσατε. Και αν όχι, τι αλλαγές θα θέλατε να γίνουν στον οργανισμό αυτόν. Για σας, για ποιος δουλεύει αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, ποια είναι η πελατεία του, ποιος εξυπηρετεί. Ναι, δουλεύω στις κάτω χώρες για το περιβάλλον. Ήταν μια από τις πιο προχωρημένες χώρες σε θέματα περιβάλλοντος και η δικιά μας εμπειρία πέρασε και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Τώρα όμω έχει αντιστραφεί αυτή η σχέση γιατί εμείς στην Ολλανδία χρειαζόμαστε σας χρειαζόμαστε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για να συνεχίσει να μας ενημερώνει και να μας βοηθάει. Πιστεύω ότι ο οργανισμός αυτός σήμερα ε, έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά του και αυτή είναι πώς να κρατήσει την Ευρώπη ενωμένη και σε αρμονία με το περιβάλλον. Και αυτό πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τα εθνικά Ινστιτούτα. Όχι μόνο με τις παραδοσιακές οντότητες, αλλά και με τις χώρες που εντάχθηκαν πιο πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλά να μάθουμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, αλλά και αυτός έχει να προχωρήσει μπροστά βάσει αναλύσεων, βάσει αξιολογήσεων και βάσει σεναρίων για το πρασίνισμα της οικονομίας, για την παραγωγή τροφίμων, πώς αυτή θα ε, συνάδει με τα συμφέροντα των αγροτών. Πολύ σημαντικό αυτό κατά τη γνώμη μου. Εκ μέρους των φιλελεύθερων, ο κύριος Γεμπράντη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χέλιγχαμπ για την παρουσίασή σας που ήταν σαφέστατη. Όντω έχετε γερή επιστημονική εμπειρία και μεγάλη εμπειρία και σε εθνικό και σε διεθνέ επίπεδο. Αυτό είναι σαφέ. Οι ερωτήσεις μου έχουν ε, απαντηθεί από εσά, τους προηγούμενους γύρους, τι προηγούμενες ερωτήσεις. Κάτι όμως έχω ακόμα να ρωτήσω. Για σας, ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Και πώς βλέπετε αυτές να αντικατοπτρίζονται στο έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Μπορεί να υπάρξει βελτίωση εκεί. Εγώ δεν βλέπω τις κύριες προκλήσεις να αντικατοπτρίζονται ακόμα στο έργο του οργανισμού. Εννοείται το κλίμα, ναι, πολύ. Και εκεί έχει να γίνει πολλή δουλειά ακόμα. Όχι για το πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα, αλλά για το ποιε είναι οι λύσεις και πώς μπορεί να αναρμονιστεί η ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά την ρήπανση του αέρος, την βιωσιμότητα, τα ενεργειακά για την Ευρώπη. Οπότε η ατζέντα για το κλίμα πρέπει να συνδυαστεί με την οικονομική ατζέντα. Αυτό βλέπω εγώ σαν μια μεγάλη πρόκληση. Και σαν δεύτερη βλέπω τη σχέση ανάμεσα στα τρόφιμα, τους πόρους, την οικονομία και το τοπίο. Πώς θα διατηρηθεί το τοπίο και δεν θα καταστραφεί στην Ευρώπη. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, αλλά αυτό βέβαια πρέπει να το συζητήσει η δικιά σας επιτροπή, ποια είναι τα αναδυόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως είναι ε, το θέμα της ρήπανση των υδάτων και των ωκεανών, πώς ε, ε, θα χρησιμοποιήσουμε τα μεγάλα βάθη και τους πόρους που βρίσκουμε εκεί σε σχέση με τη Γεωργία. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των Πρασίνων, ή Σατοχάση. Ευχαριστώ. Καθηγητά Βέλιγκτορ, από το βιογραφικό σας βλέπω ότι συμμετέχετε σε διάφορα διοικητικά συμβούλια επί του παρόντος. Ακούσαμε από τον καθηγητή Σκούλο ότι πιστεύει πως μια ενεργό δραστηριότητα στο Δυτικό Συμβούλιο σημαίνει τρεις εβδομάδε το χρόνο τουλάχιστον. Εσείς πιστεύετε ότι έχετε αυτό το χρόνο να διαθέσετε. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Κοιτάξτε, είμαι 62 ετών. θα φύγω από το πανεπιστήμιο και θα ασχοληθώ περισσότερο με το μη πανεπιστημιακό έργο. Έτσι κι αλλιώς ήδη μειώνεται πολύ η απασχόλησή μου στο Πανεπιστήμιο. Συνεπώς, το βλέπω σαν μια ευκαιρία αυτό. Τρεις εβδομάδες το χρόνο για μένα είναι κάτι απόλυτα εφικτό. Γιατί όπως σας είπα, θα μετακινηθώ κάπως από την εθνική πολιτική με την οποία ασχολούμαι στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, Γκουε, Φιντί δεν έχουν εδώ προσώπους. Και έτσι, εάν υπάρχει η επιθυμία μπορούμε να κάνουμε το περίφημο πινκ-πονγκ μεταξύ ΕΛΚ, Σοσιαλδημοκρατών, Μακέβων. Παρακαλώ, Γκουαρντίνη, όχι, δεν έχετε ερωτήσεις. Άρα, τελειώσαμε. Ευχαριστώ όλους τους εδώ παρόντες υποψηφίου, για τις απαντήσεις σας, για τις παρουσιάσεις σας, για τη διάθεση να αναλάβετε αυτό το σοβαρό καθήκον. Τώρα εμείς θα συζητήσουμε το θέμα αυτό σε επίπεδο συντονιστών για να προχωρήσουμε στην α, επιλογή. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επάνωδο. Άλλη μια πληροφορία. 6.30 όπως έχει προβλεφθεί θα γίνει συνεδρία των συντονιστών εδώ στην 4Q2. Ίσως μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα τους συντονιστές, τι λέτε, 6 και 4 τουλάχιστον, κάπως ε, νωρίτερα, τι λέτε. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Ναι, να κάνουμε μια προσπάθεια. Αν και μάλλον είναι φρούδα η ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να τους βρούμε πριν εκπνεύσει η μισή ώρα. Ας κάνει μια προσπάθεια η γραμματεία. Να αποστείλει ένα email και να ελπίξουμε ότι θα έρθουν οι συντονιστές νωρίτερα. Καλά λέει κυρία Μακέβαν, καλύτερα να τα αφήσουμε για 6.30. 6.30. Καλύτερα, να μην αλλάξουμε.